Dear I would like to start the, meeting. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Ξεκινά μία δημόσια κρέωση για από τα πλέον σημαντικά και δύσκολα ζητήματα, υποστήριξη της διαχείρισης πολιτικής συνοχής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκεί δηλαδή που είναι και η καρδιά της ανάπτυξης. Οι εμπειρογνώμονες θα μας κάνουν ε, κάποιες παρουσιάσεις και ουσιαστικά αυτοί οι πυρογνώμονε είναι και οι άνθρωποι τη πράξη σε αυτό το τομέα. Τέσσερι ομιλητέ, ε, έχουμε προσκαλέσει. Πρώτα απ' όλα την κυρία Ζιλή Πελεγκρά, διευθύντρια του Κέντρου Μηχανικών Σπουδών ε, του Μιλάνου, που είναι ένα από τα βασικά ερευνητικά κέντρα που βρίσκονται πίσω από την ε, μελέτη που έχουμε ζητήσει για τις επιχειρήσεις και έπειτα έχουμε εκπρόσωπο της Business Europe, την κυρία Μιλένα Γιαμπούρκοβα. Έπειτα έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, τον κύριο Λουκ Χάντριξ. Επίσης, θα ακούσουμε και ένα παράδειγμα από τη Σαξονία Άνχαλτ από τον κύριο Τόμας Ρίκε πολιτικό σύμβουλος στο κρατήδι της Σαξονίας Άνχελτ που θα μας μιλήσει και παρουσιάζοντας ένα case study και τη στήριξη τη μικρομεσαία επιχειρήσεις. Λοιπόν, χωρίς να μακρηγορώ περαιτέρω, θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Πελεγκρίν. Πελεγκρίν δεν είμαι σίγουρη, λέει η πρόεδρος, όπως προφέρεται το όνομά της, να μας κάνει την παρουσίασή της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω, θα σας δώσω μια πρώτη ματιά των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων ε, μιας μελέτης ε, για το κύκλο ανάπτυξης μικροπιστής επιχειρήσεων, μια μελέτη που ξεκίνησε πριν από ένα μήνα. Ε, καινούργια εντελώ τα αποτελέσματα που θα δείτε. Στόχοι τη μελέτη είναι να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε κρίσιμα ζητήματα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και για τους οργανισμούς υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι δικαιούχοι από τα Ταμεία Περιφερειακής ανάπτυξη και Συνοχής μέσω των επιλεγμένων προγραμμάτων κλειδιά και η αισθήση μα αφορά τα διευθυντικά ταμεία κατά κύριο λόγο η αναμενόμενη προσθέμενη αξία αυτής της έκθεσης είναι, μάλλον της μελέτης, είναι να μην μας δώσει έναν απλό κατάλογο θεμάτων, αλλά να γίνει μια ιεράρχηση, μια κατηγοριοποίηση των θεμάτων, μπαίνοντας σε κάποιες λεπτομέρειες για κάθε πρόγραμμα και ε, για κάθε φάση διαχείρισης των project. Στόχος είναι να εντοπίσουμε τα ζητήματα εκείνα που είναι πλέον κρίσιμη σημασία για να καταλήξουμε σε μία λίστα προτεραιοτήτων όπου θεωρείται ότι χρειάζεται περισσότερη ανάληψη δράσης. Το άλλο βασικό και ενδιαφέρον χαρακτηριστικό τη μελέτη είναι ότι συμπεριλαμβάνει του δικαιούχου, μικρομεσαίες επιχειρήσει ω δικαιούχοι, όπως και ε, φορεί υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοί ω δικαιούχοι, αλλά και ως ε, ενδιάμεση, καθώ μπορεί να έχουν ε, καθοριστικό ρόλο εν προκειμένου. Λίγα λόγια για την μέθοδο που ακολουθήσαμε ε, σε αυτή τη μελέτη. Ξεκάθαρη μελέτη σε τρεις φάσεις. Πρώτα απ' όλα αναλυτικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη είναι την τόσο πλούσια βιβλιογραφία που υπάρχει για να δούμε ποια είναι τα εμπόδια στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων. Εντοπισμός των πληροφοριών που μας λείπουν θα καλυφθούν με τη συλλογή δεδομένων. Πρώτα απ' όλα, η συλλογή δεδομένων έγινε με μελέτη περιπτώσεων από έξι επικοινωνιακά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω ε, εστιάζοντας στο κάθε επίπεδο ε, του προγράμματος που έτρεχε εκείνη τη στιγμή και εστιάζοντας σε συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό βεβαίως ολοκληρωθεί με μια ηλεκτρονική μελέτη για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα στοχεύει κυρίως στους φορείς υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον στόχο να επιτύχουμε τουλάχιστον 50 απαντήσεις. Τέλος, τα τελευταία βήματα, σύνθεση και επικύρωση των αποτελεσμάτων, βάζοντας ιδίως τα πορίσματα στο ευρύτερο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας με τον κανονισμό δηλαδή περιφερειακής πολιτικής. Όπως ε, σας ανέφερα ακροθυγώς νωρίτερα, είναι πλούσια η βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά τα εμπόδια στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Εδώ βλέπετε, αν θέλετε, μία απεικόνηση των πλέον κρίσιμων ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί. Ε, με βάση μια δημόσια διαβούλευση που έγινε με βάση την πρωτοβουλία ε, το Small Act for Europe. Ο κατάλογος αυτών είναι γεμάτος ε, γνωστά πράγματα. Διοικητικό και ρυθμιστικό βάρος, ε, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, φορολόγηση, έλλειψη δεξιοτήτων, πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειες, άθεμος ανταγωνισμός, εργασιακό δίκαιο κτλ. κτλ. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των πλουσίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση είναι πώς μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα. Ο στόχος είναι λοιπόν ακριβώς αυτός. Προκαταρτικά πρέπει να συμφωνήσουμε ή μάλλον να ορίσουμε το πώς νοούμε τον ε, κύκλο διαχείρισης των προγραμμάτων και των project. Εδώ εντοπίζουμε ε, γενικώ πώς τέσσερις φάσεις στον προγραμματισμό. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσει η μελέτη είναι η χαρτογράφηση των διαφερομένων φορέων που θα έχουν έναν ρόλο που δυνητικά θα έχουν ένα ρόλο στη διαδικασία ε, για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα διευθυντικά ταμεία. Εδώ προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις διάφορες κατηγορίες μικρομεσαίων και τον ρόλο των φορέων υποστήριξης μικρομεσαίων μέσα από τον κύκλο διαχείρισης των προγραμμάτων. Και κατηγοριοποιώντας αυτούς τους φορείς στήριξης, προτείνουμε τέσσερις ομάδες. Διακρίνοντας ανάμεσα στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμοί υποστήριξης των επιχειρήσεων, και οργανώσεις που υποστηρίζουν τη δικτύωση, τα clustering, τα cluster, συγγνώμη. Δημόσια και ιδιωτικοί φορείς μαζί Οι διάφορες αυτές κατηγορίες βεβαίως οργανισμών και ενώσεων έχουν και επικαλύψεις ε, στις, ε, στους ρόλους τους και βεβαίως έχουν και διαφορετικά καθεστώτα και ρόλους που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτά τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της μελέτης, που είναι η ταυτοποίηση μέσω της επανεξέτησης βιβλιογραφίας, λοιπόν, των βασικών ζητημάτων που μας απασχολούν σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τα ταμεία. Ξεκινούμε από τη φάση του προγραμματισμού. Εδώ έχει πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει η ποιότητα της εταιρική σχέσης. Η διαβούλευση με τους φορείς υποστήριξης αρκεί. Η παρέμβαση αρκεί για να καλύψει ανάγκες μέσα σε επιχειρήσεις. Παράδειγμα. Μια πρόσφατη έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου καταδεικνύει ότι οι ελλείψεις στην αξιολόγηση και την αποτίμηση μάλλον των χρηματοοικονομικών προβλημάτων των κρομισμένων επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε ένα κακό, κακοσχεδιασμένο εργαλείο χρηματοδότησης. Η επόμενη φάση είναι η προετοιμασία της υλοποίησης. Εδώ χρειάζονται τεχνικές λεπτομέρειες για τους κανόνες επιλεξιμότητας όπως και ευρύτερες προσπάθειες επικοινωνίας για να προσελκυστούν project, να δημιουργηθούν ιδέες που να συνάδουν με προτεραιότητες του προγράμματος. Με αυτή την έννοια, ο ρόλος των φορέων υποστήριξης ως ε, διάβλος επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικός. Η επόμενη φάση είναι η δημιουργία γέννηση των project. Εδώ βλέπετε έναν μακροσκελή κατάλογο με διάφορα σημεία. Ξεκινούμε με το σύντομο χρονικό πλαίσιο που δίνεται για την προετοιμασία των αιτήσεων. Έπειτα βλέπετε την έλλειψη βοήθειας τουλάχιστον από δημόσιους ε, φορείς για να προετοιμαστούν οι φάκελοι υποψηφιότητας κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μια δαπανηρή διαβούλευση από ιδιώτες συμβούλους. Κάτι άλλο που εντοπίζουμε είναι υπερβολικός αριθμός εγγράφων που ζητώνται. Δηλαδή, από τη μία έχουμε υπερβολικό αριθμό τεκμηρίων που ζητώνται και δεύτερον, τη ζητώνται σε χαρτί όλα αυτά. Όλα τα χρηματογνωμικά στοιχεία που συνδέονται με την έλλειψη της των προκαταβολών στη χρηματοδότηση και επίσης το αίτημα για εγγύησης. Η μακρά περίοδος που χρειάζονται οι διαχειριστικές αρχές για να αποδεχτούν ή απορρίψουν ε, μία αίτηση ε, γύρει ζήτημα διαφάνειας, το οποίο είναι πρόβλημα από μόνο του, αλλά είναι και θέμα εικόνας. Καθώς το επηρεάζει ενδεχομένως και το ενδεχόμενο ο ετών να αποτανθεί για μια δεύτερη φορά ε, για ένα άλλο project. Έπειτα η χρήση διαφορετικών αιτήσεων και διαδικασιών για διαφορετικά προγράμματα και ταμεία και αυτό δημιουργεί δυσκολίες. Και τέλος, υπερβολική προσοχή στην ε, διοικητική συμμόρφωση και όχι τόσο ε, στην ποιότητα του project. πρόγραμμα και διαχείριση, ε, συγγνώμη, προγραμμάτων και project. Ο κατάλογος εδώ είναι μικρότερος, αλλά και πάλι ε, πυκνός. Η ανάγκη για την πρόσληψη προς το προσωπικού για να αντιμετωπιστούν οι διοικητικές απαιτήσεις. Η αίσθηση που υπάρχει ότι συνεχώς αλλάζουν οι ρυθμίσεις, αλλάζουν οι κανόνες, είναι κάτι που επηρεάζει τη στάση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ακόμα και αν η στάση και η κατεύθυνση είναι θετική, μπορεί αυτές οι αλλαγές να αξιολογούνται αρνητικά ακριβώς γιατί ε, δίνουν αβεβαιότητα. Έπειτα και πάλι το θέμα των οικονομικών, χρηματοοικονομικών στοιχείων. Μπορεί να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στις ανάγκες, τις οικονομικές ανάγκες της επιχείρησης με τον κανονικό κύκλο της χρηματοοικονομικής διαδικασίας. Έπειτα οι καθυστερήσεις, ε, τα κενά, ο ρόλος των ενδιάμεσων, είναι όλα αυτά πράγματα που, που παίζουν ρόλο για τις γνωμένες επιχειρήσεις. Άλλα χρηματοοικονομικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση, την ερμηνεία, το τι είναι επιλέξιμη δαπάνη πολλές φορές, ε, είναι συχνά ε, πρόβλημα και μεγάλο βάρος για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο αφορά τον ανεξάρτητο έλεγχο, το auditing. Θεωρείται πολλές φορές δυσανάλογο και χρονοβόρο. Η δύσκολη πρόσβαση στην τεχνική βοήθεια κτλ. είναι ένα ακόμη ζήτημα. Αυτός ο κατάλογος βεβαίως εγείρει μια σειρά ερωτήσεων. Πρώτα απ' όλα, με τη συλλογή δεδομένων θέλουμε να επιβεβαιώσουμε, να επαληθεύσουμε κατά πόσον υπάρχουν υπερεκτιμήσεις, αν υπάρχουν κενά. Αλλά κυρίως να εντοπίσουμε ποια είναι τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα. και κατά πόσο μπορούν να ομαδοποιηθούν αυτά τα ζητήματα αναφάση ε, του κύκλου προγραμματισμού. Και με άλλα λόγια, υπάρχει κάποια φάση που είναι πιο δύσκολη από κάποια άλλη στον όλο κύκλο και εκεί πρέπει να δώσουμε πιο πολλές προσπάθειες για βελτιώσεις ή το αντίθετο. Μήπως είναι θέμα τομέων, δηλαδή είναι πιο πολύ τα οικονομικά ζητήματα, τα θέματα χρηματοδότησης που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Μήπως δηλαδή τα χρηματοοικονομικά είναι τα πιο αποτρεπτικά στοιχεία στην όλη διαδικασία. Επίσης, οι περιορισμοί που έχουμε εντοπίσει, μήπως εξαρτώνται από την κατηγορία των μέτρων ή από την κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναπερίπτωση. Ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα είναι ο βαθμός στον οποίο οι τοπικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τις στάση της δημοκρατίας επιχείρησης έναντι των διεθνικών ταμείων. Και σε ποιο βαθμό οι εθνικές και περιφερειακές πρακτικές και κανόνες αυξάνουν περαιτέρω τον διοικητικό ε, βάρος. Και τέλος, ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις για την πρόσβαση στα διευθυντικά ταμεία πραγματικά και ποια είναι αυτά που νομίζουν ως εμπόδια οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Δηλαδή υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίε, αλλά υπάρχουν και υποκειμενικά ζητήματα. Και πάλι το το θέμα της εικόνας που συνδέεται με την χρηματοδότηση από διεθνωτικά ταμεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε άμεσα στην κυρία Γιαμπούρκοβα που εκπροσωπεί την Business Europe που ουσιαστικά είναι συνομοσποδία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Chair, thank you for... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν που με καλέσατε σε αυτή την ακρόαση. Θα ήθελα καταρχήν να σας παρουσιάσω τις απόψεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την πολιτική συνοχής εκ μέρους της Business Europe. Καταρχήν θα ήθελα να πω γιατί η Business Europe θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική η πολιτική συνοχή. Κατόπιν θα σας παρουσιάσω κάποιες απόψεις όπως τις βλέπουν τα μέλη μας, όπως ε, διαπιστώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή την πολιτική και τις επιπτώσεις και κατόπιν κάποιες συστάσεις της Business Europe όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ε, πολιτική συνοχή. Θα σας μιλήσω για την αποτελεσματικότητα και τελειώνοντας θα αναφερθώ στις τροπολογίες της Επιτροπής. Να δούμε αν είμαι ικανή να χειριστώ αυτόν τον υπολογιστή. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα σας εκπλήξω λέγοντάς σας ότι το Business Europe στηρίζει την πολιτική συνοχής. Γιατί. Καταρχήν, η πολιτική συνοχής η οποία διαμορφώνεται για τον επόμενη χρονική περίοδο Διαμορφώνονται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, κάτι που έχει άμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βεβαίως κανείς αυτό θα πρέπει να το έχει κατά νου όταν γίνονται διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κονδύλια που διαθέτει η πολιτική συνοχή να δαπανώνται με τρόπο αποτελεσματικό. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν σήμερα σε αυτή την πολιτική. Καθότι μέχρι τώρα έχουν υπονομεύσει την δυνατότητα να φτάσουμε σε αποτελέσματα. Θα θέλαμε λοιπόν να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η ενδυνάμωση, η ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Η στήριξη των επιχειρήσεων. Και αν κοιτάξει κανείς την περίοδο 2000-2006, διαπιστώνει το 70% του 1,4 εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν κατά αυτή την στους κλάδους και στους τομείς όπου υπήρχε αυτή η στήριξη. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν εδώ τις απόψεις των μελών μας. Όπως ξέρετε η Business Europe έχει 41 ομοσπονδίες μέλη, εκπροσωπεί 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις, εκ των οποίων περίπου το 90% είναι μικρομεσαίες. Βεβαίως, πρόκειται για διαφορετικού τύπου επιχειρήσεις. Τα μέλη μας ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, κατηγορίες επιχειρήσεων με πολύ διαφορετικές εμπειρίες. Παρόλα αυτά μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν κοινέ ανησυχίες και παρατηρήσεις. Χρειαζόμαστε σωστές και ακριβείς πληροφορίες, κάτι που είναι δύσκολο να ε, βρει κανείς, όπως είπε και η κυρία ε, Πελγά στην ε, παρουσίασή μου. Θα εντοπίζω κάποιες δυσκολίες όπως η δυσκολία να κατανοήσει κανείς το Τζέρεμι. Οι δυσκολίες επίσης να βρει τις σωστές διαδικασίες και κανόνες. Ανάγκη λοιπόν για αποτελεσματικότητα. Επιγόντως χρειαζόμαστε απλοποίηση, πιο εύκολη πρόσβαση σε δημοσιονομικά εργαλεία και βεβαίως Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται λαμβάνοντα υπόψη το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Όσον αφορά την απλοποίηση, ξέρω ότι η Ομοσπονδία από την Πολωνία, μέλος της Business Europe, μας έδωσε διάφορα στοιχεία για το θέμα αυτό. Πάνω από το 10% του χρόνου δαπανάτε σήμερα σε διοικητικά διοικητικές ε, ε δραστηριότητες και βλέπετε ότι 10% των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεωρούν ότι αυτό είναι υπερβολικό, δεν μπορούν να δούνε με ποιο τρόπο μπορεί να μειωθεί αυτό το γραφειοκρατικό άχθος. Γι' αυτό και στο Business Europe θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη εναρμόνιση όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας, ψηφιακές διαδικασίες, απλοποιημένοι υπολογισμοί όσον αφορά παραδείγματο χάνει κάποιες κατηγορίες κόστους και διαδικασίες ε, απλούστερες για μικρές ε, επιχειρήσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση στην χρηματοδότηση, θα επικεντρωθώ στο Τζέρεμι. Διότι αυτό το εργαλείο μας δίνει τις ε, πιο σημαντικές ευκαιρίες για μας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά μία πρόσβαση στην ε, πολιτική συνοχή και στη χρηματοδότηση, που όπως ξέρετε έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. ακριβώς επειδή το τραπεζικό σύστημα δεν είναι διατεθειμένο να στηρίξει όλα τα σχέδια των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στρεφόμαστε προς τους περιφερειακούς φορείς. Πολλές φορές βλέπουμε ότι τα προγράμματα αυτά έχουν πολύ καλές ε, αποδόσεις, ότι τα κονδύλια αυτά μπορεί να επενδυθούν και σε άλλους ε, τομείς, Βλέπετε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε πολλές πηγές χρηματοδότησης, να μην υπάρχει λοιπόν εξάρτηση από μία συγκεκριμένη πηγή μόνο και έτσι μπορούμε να πούμε ότι γίνεται και καλύτερη κατανομή του κινδύνου για τους επενδυτές. Για να γίνει κάτι τέτοιο βεβαίω χρειαζόμαστε εργαλεία απλά, καλά σχεδιασμένα και βεβαίως που να ανταποκρίνονται στις ειδικέ ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα αναφερθώ εδώ στα αποτελέσματα αυτής της, πολιτική, της πολωνικής μελέτης. Ο ρόλος των διαχειριστικών αρχών που παίρνουν αποφάσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων, καθώς και Τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων. Υπάρχουν πολλές περιφέρειες σήμερα που γνωρίζουν το πρόγραμμα Jeremy και Jessica, δεν γνωρίζουν όμως ακριβώς πώς να οργανώσουν το κομμάτι της χρηματοδότησης, πώς να ξεπεράσουν τα εμπόδια και για ποια εμπόδια ε, μιλώ εδώ, διοικητικά, γραφειοκρατικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτό το σύστημα. Πολλές φορές δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων, έτσι ώστε να λειτουργήσει το Τζέρεμι. Όσον αφορά τους ετούντες, βλέπουμε ότι πολλές φορές οι διαδικασίες είναι γραφειοκρατικές, χρονοβόρες και υπάρχουν πολύ αυστηροί όροι και προϋποθέσεις και να είναι κανείς επιλέξιμος να μπορεί να συμμετάσχει σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι λοιπόν δύσκολη η πρόσβαση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μελέτης. Τέλος, όσον αφορά το οικοσύστημα, η Business Europe θεωρεί ότι δεν αρκεί η άμεση στήριξη και ότι εδώ χρειαζόμαστε ένα γενικότερο πλαίσιο με καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των μεγάλων εταιριών. Πολλές φορές βλέπουμε ότι μια περιοχή δεν μπορεί να δώσει κίνητρα, επενδυτικά κίνητρα σε μεγάλες επιχειρήσεις ιδιαίτερα όταν μπορούν να διευρύνουν την παραγωγή, να επεκτείνουν την παραγωγή και να δημιουργήσουν νέε θέσει απασχόληση. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για μια μικρομεσαία επιχείρηση να συμμετάσχει σε μια λυσίδα παραγωγή μια περιφέρεια. Και εδώ θα σα δώσω και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Στην Τσεχία. Μια συγκεκριμένη πολιτική έδωσε κίνητρα επενδυτικά στην περιοχή της Βοημίας, στην περίοδο 2002-2008, από τις 100 νέες θέσεις απασχόλησης που χρησιμοποίησαν, 38 ε, οφείλονται σε αυτές τις άμεσες επενδύσεις και οι υπόλοιπες 62 σε αυτού του είδους την χρηματοδότηση και την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό σε 20 διαφορετικούς τομείς. 37 δημιουργήθηκαν σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας. Αυτό μας δείχνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια συμμετοχή σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, κάτι που δίνει σταθερότητα και αυξάνει τις δυνατότητες ανάπτυξης της παραγωγής, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων. Όπως μας είπε η κυρία Πελγρά πριν από λίγο, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ξεπεραστούν κάποιες ελλείψεις, αδυναμίες ως προς τη διαχείριση παραδείγματος χάρη. Την ίδια ώρα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να υπάρξουν επενδύσεις στην καινοτομία. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές οι μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζονται τις μικρομεσαίες έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην παραγωγή, στην ποιότητα των παρεχόμενων ε, υπηρεσιών. Οι μικρομεσαίες επίσης επιχειρήσεις ε, έχουν να επωφεληθούν από αυτή τη συνεργασία, αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους, τις ε, δυνατότητες, τις τεχνολογικές, τα πρότυπα τα δίκτυα και βλέπουμε ότι αυτή η ανάπτυξη γίνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι μεγάλες επιχειρήσεις την ίδια ώρα μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα αυτά στην αγορά με μεγαλύτερη ευκορία στην τοπική, ε, εθνική αλλά και διεθνή αγορά. Καταλαβαίνετε ότι μία μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να έχει καλές ε, επαφές με τους πελάτες μέσω των δικτύων αυτών και να μπορέσει να εντοπίσει τις ε, ευκαιρίες χρησιμοποιώντας τα δίκτυα διανομής και διάθεσης στην αγορά. Επίσης το θέμα της έρευνας και ανάπτυξης είναι εξαιρετικά σημαντικό αν κοιτάξουμε τη συνεργασία μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Αυτό που χρειαζόμαστε στην Business Europe, και αυτά είναι και τα συμπεράσματά μας, χρειαζόμαστε περισσότερες ε, ρυθμίσεις και κανόνες, καλύτερη εναρμόνιση, ψηφιακές διαδικασίες, εύκολες και γρήγορες προσβάσεις για μικρά προγράμματα και σχέδια. Απλοποίηση λοιπόν το άρθρο 51 υπογραμμίζει την δυνατότητα αύξησης ε, των μέσων άρθρο 3 που αναφέρεται σε πολύ συγκεκριμένες καταρτήσεις θεματικές και ποιοι μπορεί να είναι οι δικαιούχοι. Επαναλαμβάνω, σκοπός μας είναι να βελτιωθεί η δυνατότητα αύξησης της παραγωγής αλλά και απλοποίηση των διαδικασιών σε τοπικό, περιφερειακό ε, και εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά το εργαλείο που διαθέτουμε, το Jeremy, το άρθρο 3, και αυτό μας ιδιαίτερα, ενισχύει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα νέα εργαλεία, καθώς και το άρθρο 5 για τις επενδύσεις την δυνατότητα πρόσβαση σε άλλα κεφάλαια, δίνοντας προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με μεγάλη χαρά είδαμε ότι το άρθρο 3 είναι αντικείμενο κάποιων τροπολογιών, κίνητρα για επενδύσεις κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη, καθώς και την δυνατότητα για κάποια κράτη-μέλη να προσελκύσουν στοχευμένες επενδύσεις. Ελπίζουμε ότι θα γίνουν δεκτές αυτές οι τροπολογίες. Ξέρω ότι η δική σας Επιτροπή και η Πρόεδρος ε, τις υποστηρίζουν και ελπίζω ότι οι διαδικασίες αυτές θα γίνουν απλούστερες και ταχύτερες. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Δυστυχώ να πω στου υπόλοιπου ε, επόμενου δύο ομιλητέ, ότι πρέπει να συντομεύσουν για να έχουμε και χρόνο για τι ερωτήσει και απαντήσει. Κύριε Λουκ Χέντριξ, την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που μα ε, καλέσατε εδώ σήμερα σε αυτή τη δημόσια ακρόαση. Η γραμματεία σας μου ζήτησε να απαντήσω σε τρία ερωτήματα. Και αυτό ακριβώς θα προσπαθήσω να κάνω. Πρώτον, πώς οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στα ταμεία συνοχής και ποια ήταν τα κύρια εμπόδια ε, που αντιμετώπισαν μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι εδώ, γιατί όπω γνωρίζετε κατά πιθανότητα, σημαντικό σημείο των μέτρων και των δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή πολιτική Ανταφικής ε, ανάπτυξη είναι οι πολύ μικρέ, μικρές και μεσές επιχειρήσει. Ωστόσο, παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα σε ορισμένε περιφέρειες, αρκετές πηγές μας αναφέρουν ότι μόλις 2 έως 3% των μικρών επιχειρήσεων είναι δικαιούχοι. Και ουσιαστικά αποφελούνται μόνο του 1 έως 2% αυτών των πόρων, ανάλογα και με την κατάσταση που επικρατεί στο κράτος μέλος, στο οποίο ανήκουν. Αυτό το οποίο έκανε εντύπωση ε, στο παρελθόν είναι ότι ο αντίκτυπος ε, ε, των ταμείων συνοχής είναι άγνωστος προς το παρόν. Χρειαζόμαστε ανάλυση σε βάθος λοιπόν. Παρόλο που η χρηματοδότηση ανέρχονται σε αρκετά δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, δεν υπάρχει αξιολόγηση για τον συγκεκριμένο αντίκτυπο, ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις και παρότι αυτέ εκπροσωπούν το 99,9% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ποια είναι λοιπόν τα εμπόδια. Το 2010 ήδη ε, είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις και τις είχαμε στείλει και στην Επιτροπή σας. Είχαμε κάνει μια ε, μελέτη με προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, βασιζόμενη στην εμπειρία στις ε, περιφέρειες, σε 17 κράτη-μέλη, όπου αναλύαμε τις καλές και κακές εμπειρίες που είχαμε συγκεντρώσει από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εκεί είχαμε προτείνει 105 μέτρα απλούστευσης, σε αυτές τις περιοχές. Γενικά προβλήματα, διοικητικό άχθος, οικονομική διαχείριση, έλεγχη, οικονομική έλεγχη, καθυστέρηση πληρωμών, ο ρόλος των ενδιάμεσων ε, ε, οργανισμών και διάφορα άλλα προβλήματα. Τα προβλήματα που πάνω κάτω που ανέφερε και η κυρία Πελεγκρίν. Έτσι έχετε συντομία τα βασικά εμπόδια Είχαμε λοιπόν αυτές τις 105 προτάσεις το 2010 και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που η Επιτροπή προσφάτως ε, συμπεριέλαβε στην πρότασή της αρκετές από αυτές τις ιδέες. Το δεύτερο ερώτημα που μετέθη ήταν ποια αμαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την εμπειρία. Τέσσερα είναι τα διδάγματα αυτά λοιπόν. Πρώτον, όλες οι περιφέρειες που έχουν ε, καταφέρει να εισαγάγουν αποτελεσματικά μέτρα για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι περιφέρειες που εξ αρχής έχουν συστήσει μια ε, εταιρική σχέση, μια τέτοιου είδους διακυβέρνηση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να προσδιορίσουν τις βασικές προτεραιότητες τους. Δεύτερο μάθημα, το ακριβώς αντίθετο. Οι περιφέρειες που δεν είναι τόσο δραστήριες ή δεν είναι και καθόλου δραστήριες με τις μικροπιστές επιχειρήσεις είναι αυτές που, έχουν, που δεν έχουν τέτοια εταιρική σχέση. Και αυτό για να αναλύσουμε το άρθρο 5 του ε, κοινού στρατηγικού πλαισίου που αναφέρεται στη συμμετοχή ε, των κοινωνικών εταίρων που είναι θεμελιώδους σημασία σήμερα για μας. Ε, πολλές φορές αποκλείονται de facto οι μικρές επιχειρήσεις. Αντιμέτωπες αυτές τις δυσκολίες... οι μικρέ και μεσές επιχειρήσει διστάζουν όλο και περισσότερο να αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια και υπάρχει ο κίνδυνος όλο και περισσότερες ε, μικρομεσές επιχειρήσεις και οι εκπρόσωποι του να μην θέλουν να συμμετάσχουν πλέον στα διαφορετικά ταμεία και να προτιμήσουν να συνεργάζονται με τα ίδια τα προγράμματα των περιφερειών. Και τέταρτο μάθημα και μήνυμα, συμπέρασμα θέλετε, σημαντικό για το μέλλον, Καθίστε το λένε και πιο σαφές ε, ότι οι βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 θα υλοποιηθούν σε επίπεδο περιφερειών. Και έτσι θα πρόκειται πραγματικά για μια περιφερειακή πολιτική μόνο μια, στο πλαίσιο μιας τέτοια πολιτικής λοιπόν θα μπορέσουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις να υλοποιήσουν ε, τους στόχους ε, της ε, στρατηγικής του 2020. Μετά, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα διαθέτικα ταμεία. Όπως είπα, η Επιτροπή έχει ήδη λάβει υπόψη πολλές από τις προτάσεις μας σε αυτό το τομέα. Οι βασικές ανησυχίες να τις επαναλάβω. Υπάρχει ανάγκη αποσαφήνισης ε, και του ευρωπαϊκού κειμένου και του ε, επεξηγηματικού κειμένου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για να, να αποφευθούν οι επιμέρους ερμηνείες που στο παρελθόν έχουν οδηγήσει σε, στην επικράτηση διαφορετικών ενιών ε, από ότι ε, στο αρχικό κείμενο και αυτό πολλές φορές κατέληξε σε άρνηση ε, των, τοπικών αρχών να αποδεχθούν τα προγράμματα. Ε, και αυτό σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ε, τυπικών εγγράφων που απαιτούνται. Πρέπει να υπάρχει ένα κείμενο που θα αναφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και βάσει και της ε, αρχής only once, μόνο άπαξ ε, του Small Business Act. Αυτό δηλαδή πρέπει να γίνεται μια φορά για κάθε ε, πρόγραμμα. Με ηλεκτρονική διαβίβαση των εγγράφων, ηλεκτρονική αρχιοθέτηση των εγγράφων και εναρμόνιση των δεδομένων που απαιτούνται από τα διάφορα προγράμματα. Τρίτη πρόταση, πρέπει να προσαρμόσουμε τις ε, για τις προπληρωμέ, τι προκαταβολέ, ε, Να τα προσαρμόσουμε αυτά λοιπόν στην πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό αφορά και την υλοποίηση τη αρχή τη Αναλογικότητα, που είναι μία από τι βασικέ αρχέ ε, του Small Business Act. Αυτή τη στιγμή οι ίδιες κανόνες ισχύουν ε, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή των οικονομικών δυνατοτήτων τη επιχείρηση, του οργανισμού ή του project manager. Αυτό λοιπόν έρχεται σε αντίθεση με το Think Small First, που είναι μία από τις βασικές αρχές του Small Business Act. Στο παρελθόν, αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένες περιφέρειες να στηρίζουν τα μεγάλα προγράμματα μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης χρειαζόμαστε ε, απλούστευση και ευελιξία στο έργο των ε, διαμεσολαβητών, των μεσαζόντων αν θέλετε, για τις μικροψηφίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για μικρομεσαία προγράμματα, projects. Πρέπει να δίνονται τέτοια γενικά κονδύλια για να διασφαλίσουμε την καλύτερη πρόσβαση σε τέτοιους πόρους και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους βιοτέχνες. Εμείς προτείνουμε τα ευρωπαϊκά όργανα να εισαγάγουν πέντε μέτρα. Σύμφωνα με την φιλοσοφία πίσω από το Small Business Act και των προτεραιοτήτων της. Πρώτον, να διαδραματίζουν το ρόλο του, της ενδιάμεσης αυτής ε, οργάνωσης. Η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σαφές ότι ποτέ δεν θα έχουν την ικανότητα να, να προτείνουν ή να συμμετάσχουν άμεσα σε ένα σε ένα πρόγραμμα. Από την άλλη, με τη χρήση των αυτών των ε, διαμεσολαβητών, ε, ωφελείται μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να τους καλέσουμε να, να, συμμετάσχουν σε θελοντική βάση για να ε, βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να απλουστεύσουν το έργο τους με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών ταυτόχρονα και με την διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε αυτά τα κονδύλια. Δεύτερον, πρέπει να προσαρμόσουμε τους ε, κανόνες της τεχνικής αρρωγής. Παρά την αποδοτικότητα της τεχνικής αρρωγής, λίγες είναι οι επιχειρήσεις, οι οργανώσεις επιχειρήσεων ε, που έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Και αυτό αναφέρθηκε στην μελέτη της κυρίας Πελεγκρίν. Η τεχνική αρρωγή θα μπορούσε να είναι από τα πιο αποδοτικά ε, μέσα για την καλύτερη διαχείριση σε επίπεδο εταιρική και θα διευκόλυνε και το έργο των οργανώσεων ε, επιχειρήσεων. Τρίτο μέτρο, πρέπει η Επιτροπή να συστήσει μια, ε, ένα κοινό πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης για αυτούς τους φορείς. Ο project manager δεν έχει πάντα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στη διάθεσή του και αφετέρου η συνεργασία μεταξύ του project manager και των εθνικών και εδαφικών ή τοπικών αν θέλετε διοικητικών αρχών πολλές φορές είναι ανεπαρκής ή και ανύπαρκτη. Και αυτό και έτσι διακυβεύεται η ποιότητα ε, της υλοποίησης του προγράμματος. Επομένως πρέπει να υπάρχει ε, ένα τέτοιο πληροφοριακό πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το once only, αυτή την αρχή. Λόγω της κατάστασης σε, ε, σε επιμέρους κράτη-μέλη και περιφέρειες, οι οργανώσεις επιχειρήσεων αρκετές φορές τουλάχιστον αποθαρρύνονται γιατί ε, πρέπει να δαπανούν χρόνο και χρήματα για επιμέρους διαδικασίες. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα της μελέτης. Και με αυτή, τη only once, αυτή την αρχή πρέπει να έχουμε ένα, ένα ενιαίο φορέα ε, ελεγχούν με έναν φάκελο που θα είναι διαθέσιμος για όλες τις ε, διοικητικές υπηρεσίες, τις οποίες εμείς ε, ενσωματώνουμε σε ένα σύστημα, με όλα τα απαραίτητα για όλους τους τύπους ε, ελέγχων σε όλα τα επίπεδα. Και τέλος πρέπει να ε, διαμορφώσουμε, να συστήσουμε ένα σύστημα διαμεσολάβησης για να επιλύσουμε τα ζητήματα διαφορετικών ερμηνεών που παρατηρούνται η πλειοψηφία των προβλημάτων ανακύπτει από τις διαφορετικές ερμηνείες ε, των ευρωπαϊκών, περιφερειακών ή εθνικών ε, ε, νομοθετημάτων για τις επιλέξιμες δραστηριότητε, για τους ελέγχους πληρωμών, για τους οικονομικούς ελέγχους και το καθεξής. Όλα αυτά μπορούν να επιληθούν εύκολα μέσω διαλόγου. Και έτσι θα πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο ουδέτερο σύστημα διαμεσολάβησης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρίκε, σύμβουλος πολιτικής, προσωπώντας ε, την, το τη της Σαξονίας ε, Αλχάλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας παρουσιάσει συμβολή των ταμείων για την πρόθεση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρακαλώ, θα γίνεται πιο σύντομος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πρόσκληση. Καλή σας ημέρα. Ήδη είπαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα οι προηγούμενοι ομιλητέ. Εγώ λοιπόν στη δική μου παρουσίαση θα είμαι πολύ πιο σύντομο για να μείνει και χρόνο για την συζήτηση. Θα ήθελα σύντομα να σας δείξω την περιοχή μας. Είναι ένα από τα πέντε καινούρια κρατήδια, 2,3 εκατομμύρια κατοίκους έχει το κρατήδιο αυτό. Η Μαγδεμπούργη είναι η σημαντικότερη πόλη, η πρωτεύουσα και πρόκειται για μια περιοχή η οποία παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από την βιομηχανία στον τομέα της χημίας κυρίως. 99% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. 86% των απασχολούμενων εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο κρατήδιο αυτό. Και το 61% του όλου κύκλου εργασιών, όλης της περιοχής, όλου του κρατηδίου, εξαρτάται και απορρέει από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η, ε, ο κλάδος αυτός στην περιοχή μας συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στο ΑΕΠ, στην απασχόληση βεβαίως, αλλά και στη δυνατότητα καινοτομίας της, δυνατότητες καινοτομίας της περιοχής. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθούμε εδώ στην περιοχή μας, στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Και στην σύγκριση των δικών μα δικών επιδόσεων με τις πιο ανεπτυγμένες και πιο σύγχρονες περιοχές της Ευρώπης. Γι' αυτό και η χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής ήταν εξαιρετικά σημαντική για μας. Το ξεκίνησε στη δεκαετία του 90 και την ίδια ώρα μπορέσαμε να ξεκινήσουμε μεγάλες ε, μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη της ε, περιοχής μας με τη βοήθεια των ταμείων και μετά κονδύλια που διαθέταμε, αλλά και με εμπειρογνώμονες ειδικού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για να αντιμετωπίσουμε σοβαρά κοινωνικά φαινόμενα όπως την εγκατάλειψη κάποιων περιοχών από τους κατοίκους τους. Εδώ μπορείτε να δείτε πολύ συγκεκριμένα την στήριξη για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της στήριξης της ανταγωνιστικότητας ε, των επιχειρήσεων και βεβαίως ε, η ενίσχυση της δυνατότητας καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάτι που πραγματικά αποκτά όλο και περισσότερη σημασία. Τρίτον, η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή ουσιαστικά η δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Οι πρώτοι αυτοί οι στόχοι καλύπτονται από την χρηματοδότηση και υπάρχει και ένας τέταρτος στόχος που είναι η κατάρτιση, η επαγγελματική κατάρτιση και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Εδώ βλέπετε την δομή και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ε, στην ε, περιοχή μας. Έχουμε ένα πολύ δυνατό βιομηχανικό τομέα, μίλησα για το τομέα της χημίας και βεβαίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομάζα και βεβαίως πολύ σημαντικός τομέας βιοτεχνολογίας. Ποια είναι τα πιο σημαντικά ε, σημεία για μας για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταρχήν, η στήριξη μέσω της χρηματοδότησης, οι επενδύσεις Δεύτερον, η κατάκτηση νέων αγορών. Αυτό γίνεται με την στήριξη της διεθνούς πολιτικής και στρατηγικής των επιχειρήσεών μας και βεβαίως, τρίτο σημείο, η στήριξη της ανάπτυξης των ε, επιχειρήσεων και εδώ βεβαίως θα αναφερθώ ιδιαίτερα στην έρευνα, στην καινοτομία, τα δίκτυα επιχειρήσεων με κέντρα ερευνητικά, με πανεπιστήμια κτλ. Σε αυτό το πίνακα μπορείτε να δείτε κάποια μεγέθη στο παρελθόν μέσω των ε, περιφερειακών ε, ευρωπαϊκών ταμείων στηρίξαμε κάποιους περιφερειακούς φορείς και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα για τη δεκαετία 2000-2010. Βλέπετε τα ποσά, περίπου τα 50% της χρηματοδότησης αφορούσε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην τρίτη σειρά βλέπετε τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Βελτίωση των περιφερειακών δομών και βλέπετε πολύ συγκεκριμένους αριθμούς για την προηγούμενη δεκαετία, 71 νέες θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν και σταθεροποιήθηκαν και βλέπετε τα ποσοστά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικά. Η ενίσχυση, όπως ξέρετε, της ανταγωνιστικότητας βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εδώ έχουμε τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης ενός ερωτηματολόγιου Όσον αφορά τη διαχείριση των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ερώτηση ήταν γιατί δεν είναι ανωτόμος ένας τομέας, μια επιχείρηση. 43% για λείπει εσωτερική χρηματοδότηση, 37% για λείπει εξωτερική χρηματοδότηση και 29% έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένου. Βλέπετε λοιπόν εδώ για ποιο λόγο αποφασίσαμε να στοχεύσουμε ακριβώς αυτόν τον τομέα. Ενίσχυση της καινοτομίας 2007-2011. Βλέπετε στο κρατήδιο της Αξιονίας Άνχαλ 300 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της καινοτομίας ε, στην περιοχή μας. Και εδώ σας δίνω και ένα παράδειγμα ενός προγράμματος για την στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά την σύμβαση ερευνητικών την σύναψη ερευνητικών ε, συμβολέων συμβάσεων με ταξί πανεπιστημίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν να ενισχυθεί ακριβώς ο τομέας αυτός και να προσελκυθούν εμπειρογνώμονες ειδικοί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δημιουργία δικτύων Εδώ βλέπετε στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αυτοματοποίηση διαδικασιών. Εδώ τα διαρθρωτικά ταμεία στήριξαν αυτό το πρόγραμμα και βεβαίως ένα τρίτο πολύ σημαντικό σημείο είναι η δημιουργία και η στήριξη ενός ε, τεχνολογικού πάρκου, ερευνητικών τεχνολογικών κέντρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την ε, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολύ σημαντικός ε, ρόλος και για την κατάρτιση, αυτή καθεαυτή, την επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και την ε, επανακατάρτιση υπάρχοντος προσωπικού, αλλά πολύ σημαντικό τομέας είναι και η δημιουργία νέων τομέων και η πρόσληψη προσωπικού. Την ε, δεκαετία του 90 γνωρίσαμε ένα πολύ μαζικό φαινόμενο, την μετατόπιση πληθυσμών την εγκατάλειψη κάποιων περιοχών, ιδιαίτερα της Ανατολικής ε, Γερμανίας. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια αντίστροφη, αν θέλετε, ε, τάση. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε εμπειρογνώμονες. Και εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα, το σχέδιο PFIF. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε μέσω ενός ε, φορέα, ενός οργανισμού, με τη στήριξη βεβαίως ε, του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ, αλλά και των ε, Ευρωπαϊκών Ταμείων για την προσέλκυση εμπειρογνωμόνων, την κατάρτιση ή επανακατάρτιση προσωπικού, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε κάποια κενά στην αγορά εργασίας και να εμποδίσουμε την ε, απομάκρυνση εμπειρογνωμόνων ειδικών από την περιοχή μας, είτε να προσελκύσουμε ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει την περιοχή ή που θέλουν ε, να έρθουν να εγκατασταθούν ε, στην περιοχή μας. Ποιος μπορεί να υποφεληθεί από το ΠΦΙΦ, κυρίως οι ίδιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι. Εδώ βλέπετε κάποιες μελλοντικές προκλήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως βλέπετε, πρώτη θέση στον κατάλογο έχει η καινοτομία. Πιστεύουμε ότι πραγματικά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, τη δημιουργία δικτύων μεταξύ του κόσμου της επιστήμης, της έρευνας και των πανεπιστημιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η μεταφορά τεχνολογίας και η προσέλκυση νέων ειδικών. Δύο, ανταγωνιστικότητα, στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής, αλλά και η διεθνή στρατηγική, καθώς και η κατάρτιση των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι αυτές είναι οι νέες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η χρηματοδότηση. Πολύ σημαντικός τομέας είναι και η κατάρτιση για να αποφύγουμε εγκατάλειψη και περαιτέρω έλλειψη ειδικών στην περιοχή μας. Είμαι στη διάθεσή σας για την απάντηση ερωτήσεων, αλλά μπορώ να σας δώσω και την παρουσίασή μου ε, εάν σας ενδιαφέρει με γραπτή μορφή. Σας ευχαριστώ. Ε, I would like to thank you, Mr. Να σας ευχαριστήσω κύριε Ρίκε. 15 λεπτά έχουμε στη διαθέσή μας για ερωτήσεις από τα μέλη και σχόλια, αν το επιθυμεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Νίλσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Είναι πολύ σημαντικό που γίνεται αυτή η συζήτηση αυτή τη χρονική στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια αποτίμηση του πώς έχει λειτουργήσει ως σήμερα η πολιτική συνοχή στα πλαίσια της υποστήριξης των κρεμασιών επιχειρήσεων. Εγώ μιλώ για τη δική μου εμπειρία. ήθελα πιο πολύ να απευθύνω κάποια ερωτήματα στην εκπρόσωπο της Business Europe. Εγώ προερχόμαι από τη Βόρεια Σουηδία και γνωρίζω καλά τις επιχειρήσεις στη δική μου περιοχή. Αν ρωτήσω εκπροσώπους των επιχειρήσεων έχετε λάβει υποστήριξη από δεργαταμία θα μου πούν όχι, δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν ε, μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη προβολή αυτού του έργου ρωτώ, τι πλατφόρμες έχετε για να μπορέσετε να προωθήσετε καλύτερα και να γνωστοποιήσετε τις δραστηριότητές σας στις επιχειρήσεις σε όλα τα μέρη της Ευρώπης. Έπειτα κάτι άλλο για την Business Europe και πιστεύω ότι όσοι με ακούν θα συμφωνήσουν μαζί μου. Σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί Ξέρετε, πολύ συχνά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν χρόνο για να μπουν στην διαδικασία να κάνουν αίτηση και να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδου πλατφόρμες επιχειρηματικότητας. Ε, έχουν μια πολύ πιο δύσκολη καθημερινότητα. Άρα λοιπόν, πώς θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερες πλατφόρμες, πώς θα μπορούσε επίσης Europe να βοηθήσει, να δώσει κίνητρα ώστε να αναλάβουν πιο ενεργητικό ρόλο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Yes, uh, Kelly, Η ε, Κέλλη θέλει να θέσει κάποια ερώτηση. Yes, thank you very much. Ο κύριος Κέλλη, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις. για τη συνολική συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, σίγουρα είναι σε έναν βαθμό απογοητευτική. Αλλά είναι και κατανοητή αυτή η κατάσταση γιατί συνήθως είναι τόσο μικρές αυτές οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αφιερώσουν χρόνο ε, και ανθρώπινους πόρους για να υποβάλουν αιτήσει να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύσκολα ε, πολλές φορές μπορούν να ισοσκελής του προπολογισμού τους ώστε όταν έχουν τόσο ζωτικά θέματα να του απασχολούν κάθε μέρα, δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν σε τέτοια ζητήματα. Είναι πολυτέλεια, αν θέλετε. Κάτι άλλο, βεβαίω, που θα μπορούσε να τι βοηθήσει ιδιαίτερα στι επιχειρήσει είναι τα μέτρα απλοποίηση ε, που ακούστηκε από κάποιον ομιλητή. Είπατε 105 μέτρα απλοποίησης ε, αναφέρατε. Μα για να είναι τόσο πολλά τα μέτρα απλοποίησης, ρωτώ πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση, πόση γραφειοκρατία έχει συσσωρευτεί. Δηλαδή, αν βυρίσει έναν άνθρωπο στο δρόμο και του πει, ξέρετε, έχουμε καταλήξει 105 μέτρα απλοποίησης, τι θα καταλάβει, θα σοκαριστεί. Θα δυσκολευτεί να καταλάβει την κατάσταση. Μα γιατί χρειάζονται τόσα πολλά μέτρα για να απλοποιήσουμε κάτι. Και μόνο που τα ακούς, μπερδεύεσαι. Βεβαίω, είναι ενθαρρυντικό το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είπε και ο Ρίο Ανρίκ, ότι ε, το δέχεται αυτό, να στερνίζεται και προσπαθεί να απλοποιήσει τα πράγματα. Επίση, αυτό το Think Small First ε, είναι το σλόγγαν, αλλά καλύτερα να γίνει Think Simple First. Ε, να σκεφτόμαστε απλά πρώτα απ' όλα. Ίσως έτσι να μπορούσαμε να δράξουμε πιο πολλούς καρπούς για τις μικροπιστές επιχειρήσεις διότι πράγματι είναι η ρεχοκοκαλιά της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Αν το κάνουμε αυτό, πώς θα έχουμε την ύφεση, πώς πραγματικά θα βγούμε αυτό το φαύλο κύκλο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ο κύριος Ντανικέλης. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Εν μέρη το ερώτημά μου ε, το πρόλαβαν άλλοι. Αλλά θέλω να επανέλθω και να το ξαναθέσω. Όταν σκέφτομαι την πολιτική συνοχής και πώς συνδέεται με τον ιστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φρονώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, πρόβλημα που συζητούμε χρόνια που δυστυχώς όμως δεν έχει βρεθεί λύση γι' αυτό. Ελπίζω, αν και γενικά δεν είμαι φύση αισιόδοξο, ε, στην επόμενη προγραμματική περίοδο να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε τις κατάλληλες απαραίτητες συνθήκες ώστε να είναι πιο εύκολη η προσβασιμότητα στην χρηματοδότηση και τις γνωμές επιχειρήσεις. Γιατί παραμένει αυτή η απόσταση, παραμένει αυτή η δυσκολία και είναι μια σοβαρότητη δυσκολία. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μέτρα και ρυθμίσεις τέτοιες που να στοχεύουν τον ε, ιστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ιταλία. Λέμε ότι το μικρό είναι ωραίο. Ναι, το μικρό είναι όμορφο, αλλά έχει και δυσκολίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Ενώ κάποια παραδείγματα ήδη ακούστηκαν στην συζήτηση. Φερρυπίν, ε, το θέμα της απλοποίησης, της άρσης γραφειοκρατίας, το θέμα των χρόνων είναι πολύ σημαντικό, διότι π.χ. ο χρόνος για μια επιχείρηση δεν είναι ο, χρόν, ο ίδιος χρόνος με τη δημόσια δίκηση. Η χρόνη που ακολουθεί η δημόσια δίκηση είναι πολύ μακρόσυρτη. Οι χρόνοι όμως που πιέζουν μια μικρομεσαία επιχειρήση είναι διαφορετικοί, είναι γοργοί ρυθμοί. Διότι ένα project, μια ιδέα σήμερα που θα μετα μετά από 5-6 χρόνια, ε, ε, ε, ο κίνδυνος είναι ότι αυτή η καλή ιδέα μετά από 5-6 χρόνια δεν έχει θέση στην αγορά. Δεν είναι ανταγωνιστικό το προϊόν πλέον. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, πώς θα προωθήσουμε τις διαδικασίες ε, δικτύωσης και ομαδοποίησης των μικρών επιχειρήσεων. Ακριβώς επειδή είναι πολύ μικρές, πρέπει να λειτουργήσουν από κοινού ως ομάδες. Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις. Και επειδή η ισχύ είναι εν τη ενώση, σίγουρα πολλέ μαζί μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα του πόρου. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια πραγματικά τραγική κρίση. Η κρίση βαρύνει κυρίω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Διότι είναι αυτέ που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα. Αυτέ οι επιχειρήσει έχουν προβλήματα ρευστότητα, πρόσβαση σε δανεισμό, κινδυνεύουν με πτώχευση στη σημερινή πραγματικότητα. Στην Ιταλία, αν πτωχεύσει ο ιστό μικρομεσαίε επιχειρήσει, πτωχεύει η χώρα. Ο στόχος λοιπόν αυτός είναι πρωτεύων. Πάντοτε υπό το πρίσμα της πολιτικής συνοχής. Γιατί, για έναν πολύ απλό λόγο και υπόθηκε σε μία από τις ε, παρεμβάσεις των ομιλητών. Αυτή η πόρη είναι η μόνη σίγουρη διαθέσιμη πόρη για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Οπότε, ή δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι μικροπιστέ επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους για την ανάπτυξή τους, για την καινοτομία, για τις θέσεις εργασίας ή η δυσκολία τελικά θα αποτελέσει κάτι πολύ σοβαρό και πραγματικά βαρύνει τις επιχειρήσεις αυτές. Χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και θα πρέπει να επιτραπεί στις περιφέρειες, διότι οι περιφέρειες δουλεύουν με τις προκήρυξεις διαγωνισμών και άρα κρίνουν και την πρόσβαση χρηματοδότηση. Άρα οι περιφέρειες που έχουν λόγο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την πρόσβαση αυτούς τους σπόρους. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε. Κύριε Βλάσσα, αλλά σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις γιατί αποτέλεσαν πηγαίνουν και για μας. Και θα ήθελα να πω ότι όλοι αυτοί οι στόχοι, οι παρατηρήσεις, οι απόψεις θα μπορούσαν να ενταχθούν ε, σε σχέδια νέων νομοθετημάτων. Όμως ε, εκφράζεται η ανάγκη καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ε, επιχειρηματιών και τη δημόσια διοίκηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η απλοποίηση, η πιο εύκολη πρόσβαση στι δημόσιε προμήθειε και άλλα τέτοια στοιχεία. Γι' αυτό η συμμετοχή των εκπροσώπων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι απαραίτητη σε αυτή τη συζήτηση. Έχετε και εσεί την ίδια άποψη. Ευχαριστώ. Ε, μη Κασπινής Ευχαριστώ. Αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για τις ε, παρουσιάσεις σας. Αντικατοπτρίζουν με πολύ καλό τρόπο τις ε, προτεραιότητες, ε, τα εμπόδια και κάποια από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να υπερπαιδηθούν αυτά τα εμπόδια. Πράγματι, μαζί με την Επιτροπή καταφέραμε να βελτιώσουμε κατά κάποιον τρόπο την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολλά όμως μένουν ακόμα να γίνουν σε ό,τι αφορά την γραφειοκρατία, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την απλοποίηση αυτής της πρόσβασης και της βελτίωσης της πρόσβασης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στις ευρωπαϊκές αγορές, γιατί υπάρχει και τέτοια ανάγκη. Αναφέρατε κάποιες προτεραιότητες όπως ε, η απλοποίηση των κανόνων, η ευκολότερη χρηματοδότηση και βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά. Έχοντας κατά νου όλες τις τρυπολογίες που έχουμε ήδη υποβάλει στην Περιφερειακή Πολιτική ε, Επιτροπή αλλά και σε άλλες επιτροπές, θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας για το εξή θέμα. Πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να απλοποιήσουμε την διασενιωριακή κάλυψη των χρεών και, και τι σημαίνει με την νομική βεβαιότητα για αυτή την ε, αποκατάσταση του χρέους ε, και τι θα γίνει με την οδηγία των καθυστερημένων ε, πληρωμών που προβλέπεται μόλις για τον Ιανουάριο του 2013. Ναι, ο συνάδελφος ε, Βλάσακ σας ε, ζήτησε και περαιτέρω εξηγήσεις σε ό,τι αφορά την ε, πιο εύκολη συμμετοχή στους δημόσιους διαγωνισμούς. Αυτά τα ερωτήματά μου. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να συνεργαστούμε και στο μέλλον όπως συνεργαζόμαστε τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Thanks. Mr. please. Yes. Ευχαριστούμε κύριε Σόλμπρεχτε. Ευχαριστώ πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Είναι πολύ σεξι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τελευταία. Είναι ένα αγαπημένο θέμα πια. Αλλά δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε, πια, να παλέψουμε για τις μικρομεσαίες. Όλοι ε, επιθυμούν την συμμετοχή τους. Κανένας δεν έρχεται σε αντίθεση, δεν διαφωνεί με την ε, με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ω μία από τις τρεις βασικές προτεραιότητε. Το δικό μου ερώτημα ως προς τους συντάκτε των εκθέσεων είναι γνωρίζουμε εάν το μέγεθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το ορθό για τα 27 κρατημέλη. Ποια είναι τα όρια, ποιες θεωρούνται πολύ μικρές και ποιες θεωρούνται μικρές ή μεσές επιχειρήσεις. Στη δική μας επιτροπή ψηφίσαμε για κάτι που θα είναι επιλέξ... για το οποίο θα είναι επιλέξιμες και οι πολύ μικρές και οι μικρές και οι μεγάλες και οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Αφορά λοιπόν και με τις μεγάλες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με μικρομεσαίες. Επομένως εγώ ρωτώ, τι συμβαίνει με τον καλύτερο προσδιορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα είναι κάτι χρήσιμο. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσει πλέον γίνονται όλα και μεγαλύτερες. Στη χώρα μου είναι αρκετά μεγάλε. Και δεύτερον, οι ευρωπαϊκές διοικητικέ διαδικασίες είναι πιο δύσκολε από τις ε, τραπεζικέ, Δηλαδή, αν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, πάνε σε μια τράπεζα για να ζητήσουν χρηματοδότηση, αυτό είναι πιο εύκολο από το να στραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Γιατί εμει ε, ε, προβάλλουμε ενστάσεις, κάνουμε παράπονα, διαμαρτυρόμεθα, αλλά τι σημαίνει τελικά. Είναι απλή η διαδικασία ή όχι. Βεβαίω δεν, είναι, δεν ασχολούμαι με αυτόν τον τομέα. Αλλά και η δημόσια χρηματοδότηση δεν πρέπει να είναι και τόσο εύκολη διαδικασία, ούτε περίπλοκη ούτε υπερβολικά απλή. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλές παρατηρήσεις, ερωτήσεις θα μπορούσα να κάνω για να... γιατί πήγαμε ε, μέσω της συζήτησης και πέρα από τα θέματα που έθιξαν ε, οι ομιλητές στι παρουσιάσεις τους. Αρχικά να σας ευχαριστήσω που μας προσκαλέσατε, που αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία ε, για την διεξαγωγή αυτής της ε, μελέτης. Κάποια από τα αρχικά συμπεράσματα που ε, αναφέρθηκαν στις αρχικές παρεμβάσεις αντανακλούν και τα όσα ακούσαμε σε προηγούμενες συζητήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν. Σημείωσα ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι προφανώς θέμα θεμελιώδους σημασίας που αφορά όλες τις επιχειρήσεις, βεβαίω και τις ε, μικρομεσαίες. Με τα χαράς μπορώ να πω ότι στην πολιτική συνοχή δίνουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό το θέμα Αναφέρθηκε και η θεματική συγκέντρωση για τις ε, ε, η μελλοντική χρηματοδότηση του Ταμείου ανάπτυξη. Ανάπτυξης. Ε, σίγουρα θα υπάρξει και επαναπραγματισμός αυτού του εγχειρήματο όταν θα δίνουμε χρηματοδότηση, πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα προς τους συντάκτες της μελέτης δείξατε ένα διάγραμμα που αναφερόταν στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ακούσαμε και τις παρατηρήσεις ε, από την ε, Σαξονία Ανχάλτ. Είναι κέριο ε, αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μου πείτε τι είδους χρηματοδότησης εννοούμε εδώ. Υποτροφίες, δάνεια, ε, επενδύσεις υψηλού κινδύνου, άλλες μορφές χρηματοδότησης με, με vouchers και άλλες τέτοιες ε, επιλογές. Μετά, αυτή η χρηματοδότηση απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις ή σε ομίλους επιχειρήσεων ή σε συνεργασίες επιχειρήσεων και ερευνητικών Ινστιτούτων. Και πάλι για την ε, πρόσβαση στη χρηματοδότηση μετά. Ε, γιατί ποσά μιλάμε για μικρές χορηγίες ή υποτροφίες που εκεί θεωρώ ότι το, το να έχουμε ε, πρέπει να, να θίξουμε και το θέμα της αναλογικότητας μεταξύ του όγκου, του έργου και του χρόνου. Αλλά μιλάμε για μικρά ποσά αν μείνω στην παρατήρηση ότι μόλις 2-3% ε, των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στα διευθυντικά ταμεία, εμένα αυτό δεν με εκπλήσει. Αν ε, διαιρέσετε δια των 19 εκατομμυρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φαντάζεστε. Προφανώ και δεν μπορεί να έχει κάθε μικρομεσαία επιχείρηση πρόσβαση σε τέτοια χρηματοδότηση. Η ποσότητα ποιο είναι το ποσό της χρηματοδότησης που επιθυμούμε, γιατί αυτό καθορίζει και τα μέσα παρέμβασης που διαθέτουμε. Άλλο ερώτημα. Και βασίζομαι σε μια από τις τελευταίες παρατηρήσεις για την πρόσβαση στις δημόσιες ε, προμήθειες, ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι ανγένειες επιχειρήσεις σε περιόδους κρίσης είναι η ε, πρόσβαση στους πελάτες τους, όχι τόσο στην, σε υποτροφία. Στους φερέγγιους πελάτες, όχι τόσο στις, σε άλλα τέτοια κονδύλια. είναι μια εξάντε προϋπόθεση της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση των ε, επιχειρήσεων στην μελλοντική πολιτική συνοχής και από ό,τι έχω παρατηρήσει στις διαπραγματεύσεις δεν ε, θέλουν να συμπεριλάβουν αυτή την ε, εκ των προτέρων προϋπόθεση. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση λοιπόν. Πολλά ζητήματα υπάρχουν από αυτού. Είναι πολύ ενδιαφέρον αλλά θα επιταχύνω Περνάω στη συμμετοχή και εμπλοκή των μικρομεσών επιχειρήσεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμπεριλάβουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον ε, ορισμό των ε, προγραμμάτων, ποιες είναι οι προϋποθέσεις κτλ. Η Επιτροπή στις προτάσεις για, τη, για τα ταμεία ε, συνοχής προβλέπει ενδυνάμωση της εταιρική σχέσης και συμμετοχή των μικρομεσών επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς ε, προάγουμε ιδιαίτερως από το που ε, αναφέρθηκε πρώτη φορά το θέμα της καινοτομίας, ε, των στρατηγικών καινοτομίας και εφιούς εξειδίκευσης. Και προς τα εκεί πιέζουμε να υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση για την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών. Και τέλος, απλοποίηση. Είναι πράγματι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής. Σημείωσα τα 105 μέτρα απλοποίηση, σίγουρα θα μπορούσαν να είναι και παραπάνω. Νομίζω ο κύριος Άινστάιν αναφέρθηκε ότι το να κάνει κάποιος, ε, να περιπλέκει τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο, αλλά το να τα απλοποιεί είναι το πιο, ε, είναι πολύ εύκολο μάλλον, το να τα απλοποιεί κάποιος είναι το πολύ δύσκολο. Θέλουν περισσότερη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ε, και το καθεξής. Να χρησιμοποιούμε τέτοια μέσα ε, ηλεκτρονικά. Καλούμε τα, κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τα, τους πόρους ε, τεχνικής αρρωγής για την καλύτερη υλοποίηση των μέτρων τους, για να προαγάγουμε στα κράτη-μέλη την ιδέα ότι έχουν τον ηγετικό ρόλο για την βελτίωση της επικοινωνίας τους μεταξύ των διαφορών προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στους ε, ομιλητές μας, αλλά παρακαλώ να μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά έκαστος. Just, uh... Λοιπόν, για το πρώτο ερώτημα, για τις πλατφόρμες που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων στην χρηματοδότηση. Υπάρχουν πολλές τέτοιες πλατφόρμες ε, σε εθνικό επίπεδο. Και εδώ οι συνάδελφοι μπορούν να πούν λίγα λόγια για το πώς δουλεύουν με αυτές τις πλατφόρμες και εμεί έχουμε σχετική εμπειρία στην Business Europe όμω, το πρόβλημα τελικά ε, καταλήγει να είναι πάντοτε είναι πώς μπορεί να γνωρίσει κανείς για την ύπαρξη αυτών ε, των μορφωμάτων. Δηλαδή, θα πρέπει κανεί ηλεκτρονικά με ένα κλικ ε, να λέει θέλω να κάνω μια επιχείρηση, θέλω να βρω αυτό κτλ. Οπότε να μπορεί να παίρνει πληροφορίες, πώς μπορεί να πάρει χρηματοδότηση από διαφορετικά ταμεία, από διαφορετικούς κουμπαράδες ε, για να μπορέσει να έχει μια καλύτερη και εικόνα της κατάστασης για τις ε, προκηρύξεις διαγωνισμών. Πολύ συχνά βασίζονται στη συγχρηματοδότηση Είναι λοιπόν, και επειδή η χρηματοδότηση ε, ακολουθείται από πολύ αυστηρού κανόνε, ε, πολύ συχνά οι διαγωνισμοί είναι ένα δύσκολο πράγμα. Δεν θέλω να καταχρήσω περαιτέρω του χρόνου σα, να δώσω το λόγο στου αδέλφου. Ε, μάλιστα, ευχαριστώ πολλά τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα στον κύριο Κέλλη. Ελπίζω να μην ε, ασκήσετε κριτική σε μένα για αυτά τα 105 μέτρα. Εμεί είμαστε σοβαρή οργάνωση. Προτείνουμε 105 μέτρα Απλοποίηση. Ξέρετε, το σλόγγαν που χρησιμοποιήσατε εσείς για την απλοποίηση εν γέννη αφορά και την έξυπνη νομοθεσία, το Smart Regulation, έχει ως γνώμονα το Do Not Simplify. Μην γενικεύετε, μην απλοποιείτε τα πράγματα, μην τα υπεραπλουστεύετε. Δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει, είναι περίπλοκο. Κύριε Ντεάντζελης, είπατε ε, ότι θα πρέπει να ε, ομαδοποιηθούν, να ενωθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα υπάρχει ισχυρή παράδοση α, μιας τέτοιας κίνησης στη χώρα σας. Και έτσι απαντώ και στον κύριο Βλάσεκ. Το βασικό μήνυμα που ήθελα να περάσω εγώ είναι ότι θέλουμε διακυβέρνηση, ξεκάθαρη διακυβέρνηση των εταιρικών σχέσεων. Εταιρικών σχέσεων ανάμεσα στους δημόσιους φορείς και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το ερώτημα της κυρίας Μανέσκου για την καθυστέρηση των πληρωμών. Ε, ναι. Τώρα είναι λιγάκι αργά έχει ψηφιστεί αυτό το θέμα ήδη και γνωρίζετε ότι για αυτό το θέμα των καθυστερήσεων τα κράτη-μέλη δεν ήθελαν προτέρα εφαρμογή και μπορεί να είναι μάρτυρες και ο κύριος Ντεάντζελε ότι και στην Ιταλία πληρωμή των επιχειρήσεων ε, που πλήττονται από αυτό το πρόβλημα ε, δεν θα δουν λοιπόν ε, τους επόμενους μήνες πληρωμές. Κύριε Όλπρεχ, για τις γνωστές επιχειρήσεις μάλλον πρέπει να τα πούμε μεταξύ μας. Ξέρετε, συνήθως έχω σταματήσει να λέω στους ανθρώπους ε, ε πράγματα στις επιχειρήσεις, γιατί πράγματι μπορεί να είναι σεξι, να είναι τόσο ελκυστικές οι μικρές επιχειρήσεις, αλλά γίνεται κατάχρηση και του όρου και όσων ε, λέμε και τις χρησιμοποιούμε. Ξέρετε, ε, λέμε μικρομεσαίες, ενώ πάνω από το 95% είναι πραγματικά πολύ μικρές επιχειρήσεις με κάτω από 50 εργαζόμενους. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για ένα οικονομικό πλαίσιο στην Ευρώπη, καθώς η μέση ευρωπαϊκή εταιρεία έχει 5 υπαλλήλους, είναι πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για αυτές τις επιχειρήσεις μιλάμε και αυτές εκπροσωπούμε. Ευχαριστώ. Ich möchte im Prinzip äh, Καταρχήν θα απαντήσω σε τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, το θέμα της πλατφόρμας. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά απαραίτητο να δημιουργηθούν δίκτυα υποστήριξης, όπως ε, το δίκτυο Enterprise Europe. Να ενισχυθούν αυτά τα δίκτυα, καθότι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και στην ε, συμβουλευτική δραστηριότητα που έχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάνω να υπάρχουν αυτοί οι φορείς γιατί η μία περιοχή από την άλλη στην Ευρώπη παρουσιάζουν πολύ μεγάλες διαφορές. Ακόμα και στην ίδια μας τη χώρα, στη Γερμανία, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Στη Δυτική Ευρώπη, αν θέλετε, η μέση μεσαία επιχείρηση έχει περίπου 250 ε, άτομα εργαζόμενους, ενώ στην ε, δική μας περιοχή, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, 90. Καταλαβαίνετε ότι η χρηματοδότηση εξαρτάται λοιπόν από πολλούς παράγοντες, από τις ειδικέ ανάγκες και τα διαρθρωτικά τομεία εδώ αποτελούν, συνεχίζουν να αποτελούν μια πάρα πολύ σημαντική πηγή για μας. Βεβαίως είναι οι κανόνες όπως έχουν θεσπιστεί, αποφασιστεί και θα εφαρμοστούν από το χρόνο όπως η Βασιλεία 3 δυσκολεύουν πάρα πολύ την κατάσταση όσον αφορά την ιστροή κεφαλαίων από τον τραπεζικό τομέα στις επιχειρήσεις μας και ξέρουμε ότι θα πρέπει με κάποια μέτρα να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ιδιωτική αγορά κεφαλαίων. Πολύ σύντομα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακούσαμε και πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Και πιστεύω ότι βάσει όλων αυτών που είπαμε σήμερα θα πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία μας. Μιλήσατε για τον ορισμό των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν ξέρω αν υπάρχει μία για την κάθε χώρα ή ένας ορισμός, σε βάση περιπτώσει, για όλη την Ευρώπη. Όντως υπάρχουν μεγάλες διαφορές από τη μία περιοχή στην άλλη. Ακούσαμε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και από την Επιτροπή. Μια ανοιχτή ερώτηση. Τι τύπος χρηματοδότησης αρμόζει. Επίσης, σε τι ποσότητα. Η ποσότητα δεν είναι το μόνο κριτήριο βεβαίως. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στους ε, δημόσιους διαγωνισμούς. Και αυτό σε αντίθεση με τις επιδοτήσεις. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, επιτρέψτε μου. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση, θεωρητική θα έλεγα. Εμείς όμως μιλάμε για τα θέματα επιλεξιμότητας. Γι' αυτό και μιλούμε για τις πιο αναπτυγμένες περιοχές εκ των οποίων το 80% θα πρέπει να στοχεύουν τρεις προτεραιότητες. Και το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε ακριβώς στον τομέα αυτό, ποιοι είναι οι κανόνες επιλεξιμότητας. Όχι μόνο για τις μικρομεσαίες, αλλά και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια συζήτηση για το ποιος είναι σε αυτή την κατηγορία δεν θα αρχίσουμε θεωρητική συζήτηση. Μιλάμε όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Αυτό μας ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας. Επανερχόμαστε στο σημείο 7. Κυρία Μανέσκου. Το θέμα αφορά την γνωμοδότησή σας. Shall we wait for a few minutes or... Να περιμένουμε λίγα λεπτά. europene Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σαν σκοπό τις ε, κατευθυντήριες γραμμές, τις προτεραιότητες όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα καθώς και τα ψηφιακά δίκτυα για τις ε, τηλεπικοινωνίες. Και αυτό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Διασύνδεσης. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Επιτροπής και πιστεύω ότι θα παίξει ένα ρόλο ενίσχυσης της ανάπτυξης και θα μας επιτρέψει να πλησιάσουμε πιο κοντά στους στόχους της στρατηγικής του 2020. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι τα δίκτυα αυτά ενισχύονται και η πρόσβασή τους είναι ευκολότερη και για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τους πολίτες. Σήμερα αυτή η πρωτοβουλία θα μπορέσει να είναι χρήσιμη για όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρξει πρόσβαση ιδιαίτερα στις μειονεκτούσες περιοχές, τα τα ταμεία βεβαίως τα πλαίσια της ψηφιακής ατζέντα μας επιτρέπουν να υλοποιήσουμε τους στόχους αυτούς και παίζουν και ένα συμπληρωματικό ρόλο όσον αφορά την πρόσβαση στα δίκτυα αυτά, ιδιαίτερα σε εποχές όπου προσπαθούμε να αναπτύξουμε περισσότερα την ηλεκτρονική, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις τηλεπικοινωνίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν αξιόπιστα δίκτυα και δυνατότητες εναλλακτικές όσον αφορά κάποιες απομακρυσμένες υπαίθριες περιοχές και με αυτόν τον τρόπο και την ανάπτυξη των δικτύων αυτών θα μπορέσουμε να έχουμε όλη πρόσβαση ταχεία και αποτελεσματική. Εδώ υπάρχει ένας κατάλογος ε, προγραμμάτων, σχεδίων επιλέξιμων προς χρηματοδότηση στα πλαίσια αυτού του μηχανισμού. Χρειάζεται μια σχετική ελαστικότητα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Θα θέλαμε ιδιαίτερα να υπογραμμίσουμε τη σημασία τη συμμετοχή των τοπικών φορέων, των περιφερειακών φορέων και οργανισμών, οι οποίοι θα πρέπει να υποφεληθούν από διάφορα μέτρα στήριξης, βελτίωση της διοικητικής τους δομής, των δυνατοτήτων τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να καλύψουν τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες. Στηρίζω ιδιαίτερα την πρωτοβουλία της Επιτροπής και βεβαίως θα ζητήσω από τους συναδέλφους να υποβάλουν τροπολογίες. Ευχαριστώ. Εγώ παίρνω το λόγο εξ ονόματος του Σκιώδους, του κυρίου Ρόιλ ο οποίος μου είπε να τον ε, αντικαταστήσω. Εμείς βεβαίως ε, σαν ε, πολιτική ομάδα είμαστε υπέρ της στήριξης αυτών των μέτρων και βεβαίως θεωρούμε ότι εδώ θα πρέπει η αγορά να είναι ανοιχτή και να υπάρχει πρόσβαση για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σύμφωνα με την εισηγήτρια. Διάφορα μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προώθηση αυτού του ανοίγματο της αγοράς και την ίδια ώρα η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη είναι κάτι στο οποίο μπορεί να ενσωματωθεί όλη αυτή η πρωτοβουλία. Προγράμματα τα οποία μπορούν να υποστηριχθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία Γι' αυτό και θεωρούμε ότι η πρόταση της κυρίας Μανέσκου θα πρέπει να ενσωματωθεί σε μια γενικότερη προσπάθεια θέτοντας πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες όσον αφορά τα ψηφιακά δίκτυα και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, σε λιγότερο πύκνο κατοικημένες περιοχές και σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Τέλος, θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε αβέβαιες επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν οι επενδυτές να συνδυαστούν με τις τοπικές αρχές έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος ε, μη βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Αναμυράτα. Αναμυράντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Χρυσόγελε. Ευχαριστούμε θερμά την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση. Πρόκειται για ένα θέμα που αγγίζει τον ίδιο τον πολίτη, τον πολίτη που κύριο ζει στην Ήπεθρο, στις ορεινές και πλέον απομακρυσμένες παραμεθόρες περιοχές της Ευρώπης. Πολύ συχνά η αγορά η ίδια δεν μπορεί να κινηθεί δεν ε, μπορεί να κάνει κάτι γιατί πολλές υπηρεσίες είναι πολύ ακριβές. Π.χ. τα ευρυζωνικά δίκτυα είναι πολύ ακριβά για κάποιες περιοχές μακρινές και για αυτό το λόγο βλέπουμε να υπάρχει ένα χάσμα και να απομακρύνεται όλο και περισσότερο ο τρόπο τον οποίο κηρυθούν, τον οποίο αναπτύσσονται τα αστικά κέντρα με τι πλέον απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές βλέπουμε ότι τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στις αστικά κέντρα και την Ήπεθρο. Δεν μιλώ γενικά και όριστα, μιλώ για το δικό μου το χωριό, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από μια μεγάλη πόλη, θα έλεγα. Λοιπόν, στο χωριό μας δεν υπάρχουν ευρυζωνικά δίκτυα. Αυτό είναι ένα καθημερινό παράδειγμα που βιώνουν πολλοί άνθρωποι σε διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, διαβάσαμε το αρχικό σα κείμενο, θα κάνουμε όμω κάποιε τροπολογίε επικοδομητικέ γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να κινηθούμε όλοι από κοινού. Εν προκειμένου. Ευχαριστώ. Thank you. If there is nobody else who want... Ευχαριστώ. Αν ε, δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, παρακαλώ η κυρία Μανέσκου να απαντήσει. Αν το επιθυμεί Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τις ε, τοποθετήσεις τους. Όπως ε, ήδη είπα στην ε, πρώτη μου παρέμβαση, η διασύνδεση της Ευρώπης θα πρέπει να έχει λειτουργήσει συλλογματικά προς τα διαφορετικά ταμεία για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ολοκληρωμένα και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Βεβαίω, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε την ανταγωνιστικότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιφέρειας χωριστά. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαβούλευση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία μαζί σας. The for... Καταληκτική ημερομηνία για τροπολογία είναι η 20 Σεπτεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Προχωρούμε στο σημείο 22. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κατρίν Γκρέσ, να παρουσιάσει τη σχέδια γνωμοδότηση για τι άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξη τη κοινή γεωργική Πολιτική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Όπω ξέρετε, η μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 2014-2020 είναι ένα από τα μεγάλα διακυβεύματα της θητείας μας Στην πρότασή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τρεις μεγάλους ε, στόχους για αυτή τη ε, μεταρρύθμιση. Συγκεκριμένα, ε, βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τέλος, ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. Αυτοί οι τρεις στόχοι είναι θεμελιώδης σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη και για την Επιτροπή μας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το greening και για τη βιώσιμη ανάπτυξη δυστυχώς ε, ε, αποδυναμώθηκαν ε, κατά τη διάρκεια των μηνών, κυρίως από την πρόταση του Νοεμβρίου του 2010 και μέχρι τον Οκτώβριο του 2011. Ε, ωστόσο, η εξισορρόπηση τη ε, κοινή πολιτική είναι θεμελιώδη σημασία για την διατήρηση των θέσεων εργασία, ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη, για να μην πω και συνεκτική και βιώσιμη. Γι' αυτό σας ε, προτείνω κάποιες ε, τροπολογίες για τον κανονισμό που αφορά τις άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών που επιτρέπει την εφαρμογή μιας βιώσιμης, ε, στοχευμένης και ρεαλιστικής ε, προσέγγισης. Θα σας παρουσιάσω τις βασικές αρχές. Εκεί όπου η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλά για διαφοροποίηση των καλλιεργειών. Στο άρθρο 30. Εδώ προτείνω να κάνουμε λόγο για ε, ε, ε που ε, επιβάλλει την εκπεριτροπή καλλιέργεια τεσσάρων διαφορετικών καλλιεργειών. Αυτό θα πρέπει να γίνεται κυρίως στους ε, ε, βοσκοτόπους ε, που επιτρέπει την αύξηση των θετικών επιπτώσεων για τους γεωργούς αυξάνοντας τις γεωργικές τους επιλογές βοηθώντας τους να σταθεροποιήσουν το αγροτικό τους εισόδημα αλλά και να μειώσουν την χρήση ζυζανιοκτώνων. Αυτό θα βελτίωνε το βιωτικό επίπεδο των των κατοίκων της υπαίθρου, αλλά και θα βελτίωνε και τον ε, κοινωνικό και οικονομικό ιστό της υπαίθρου. Προτείνω επίσης να μιλάμε για οικολογικές υποδομές στο άρθρο 32, αντί για ε, επιφάνειες ή περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος ε, προκειμένου να συμπεριληφθεί και η βιοπικιλότητα, η Ε, και τέτοια στοιχεία του, του, του περιβάλλοντος ε, να συμπεριληφθούν σε αυτή την πολιτική. Γιατί αν ε, μιλήσουμε μόνο για ένα όπως υπάρχει τώρα, μιλάμε μόνο για ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εδαφών και αποκλείονται άλλες περιοχές. Αυτό θα βελτίωνε και, τις, και τα οικοσυστήματα και την διατήρηση της πεποικιλότητάς τους που είναι πολύ σημαντική για μια βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και για την ε, διατήρηση ε, της ε, εδαφικής συνοχής. Δεν θα ήταν ευταίο μόνο μερικές συγκεκριμένες ζώνες να είναι σε καλή κατάσταση. Πρέπει να υπάρχει πολιτική για το σύνολο των ευρωπαϊκών εδαφών. Μια τέτοια διάταξη ε, επιτρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών, ε, ε, της ευρωπαϊκής επικράτειας, επιτρέποντας συγκεκριμένες καλλιέργειες προσαρμοσμένες στον κάθε τόπο και στην κάθε περιφέρεια. Επίσης προτείνω να τροποποιηθεί το άρθρο 20 για να υποβληθεί σε αξιολόγηση, σε πρώτη αξιολόγηση αντικτύπου ε, κάθε αλλαγή στο σύστημα άμεσων πληρωμών σε περιφερειακό επίπεδο. Η Επιτροπή βασίζεται μόνο στα οικονομικά ή αγρονομικά χαρακτηριστικά των περιοχών, ενώ υπάρχει και το αγροτικό τους δυναμικό ή η διοικητική τους δομή. Θα ήθελα να αποφύγουμε την ε, παράταση των πληρωμών βάσει ιστορικών κριτηρίων, ε, προτείνοντας την ε, διεξαγωγή εξολόγησης αντικτύπου πέρα από αυτές που προτείνονται από την Επιτροπή. Με, κατά τον ίδιο τρόπο προτείνω να υπάρχει διαφάνεια στα αποτελέσματα των μελετών με τη δημοσίευσή τους. Άλλη τροπολογία 5 για την ε, σημασία ε, ύπαρξης ενδιαφέροντος για κάποιες ε, καλλιέργειες που σέβονται το περιβάλλον. Εδώ πέρα συγκεκριμένα αναφέρομαι στι στις ορεινές περιοχές όπου η γεωργία είναι εκτεταμένη. Η, η παραγωγή εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι ποσοτική αλλά ποιοτική. Και αυτή η συνδεδεμένη στήριξη είναι μία από τις λύσεις για να μπορέσουν ε, οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν ε, τις διάφορες προκλήσεις οικονομικές και άλλες που αντιμετωπίζουν. Αυτό το μέτρο ε, θα επιτρέψει να, την στήριξη της ποιοτική γεωργίας βάσει και της συνθήκης της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εξάλλου, αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω και τροπολογίες ε, επί της ε, βάσης ε, για την ανάπτυξη της υπαίθρου και στο πλαίσιο της μελλοντικής κοινής γεωργικής πολιτικής. Είναι θεμελιώδη σημασία να λάβουμε υπόψη σε μεγαλύτερο βαθμό τα περιφερειακά ή εδαφικά στοιχεία των περιφερειών μας. Ε, έτσι θα έχουμε μια συνεκτικότητα στη χρηματοδότησή μας ε, βάση και της νέας πολιτικής συνοχής για το 2014-2020. Μία από τις τροπολογίες μου στο άρθρο 14 λοιπόν προτείνει να δώσουμε στα κράτη-μέλη μεγαλύτερο εύρος στο ε, Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προτείνοντας μεγαλύτερο ποσοστό των εθνικών κονδυλίων να μπορεί να αφοσιωθεί, να, να πάει ε, σε αυτό το ταμείο. Εκεί που η Επιτροπή προτείνει ένα μέγιστο 10% των εθνικών κονδυλίων, εγώ προτείνω να πάμε στο 20%. Τα κάτι μελη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη, στήριξή τους ε, στην περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης, για το 14-20, με μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ε, το ε, Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα συμπεριληφθεί σε αυτήν την ε, υλοποίηση των κοινών στόχων με την συγκέντρωση πολλών πόρων. Στο ίδιο άρθρο η Επιτροπή προτείνει και το αντίθετο, δηλαδή να να ανακτήσουμε ένα ποσοστό των κονδυλίων από την περιφερειακή ανάπτυξη στις άμεσες πληρωμές. Αυτό θα ήταν ε, δυνατόν να αναφερθεί στο ίδιο άρθρο. Εγώ θέλω να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες για όλους, αλλά ε, αρνούμε να αποδεχθώ και μια μείωση των της ανάπτυξης υπαίθρου, γιατί αυτή θα είναι πολύ ε, δυσμενής για την εδαφική συνοχή, ιδίως στις, περιοχές, περιφέρειες που έχουν μεγάλο ποσοστό αγροτικών περιοχών. Στην τροπολογία 3 τέλος έχω την πρόταση της Επιτροπής των Περιφερειών όπου προτείνουμε την εφαρμογή των συμβάσεων, των εδαφικών ε, συμβάσεων με ωφέλιμες για το περιβάλλον αγροτικές πρακτικές. Ε, έτσι προτείνω να υπάρχουν εδαφικές συμβάσεις μεταξύ των περιφερειακών αρχών και των γεωργών. Αυτές οι συμβάσεις ε, θα επιτρέψουν να κάνουμε ένα μητρό, αν θέλετε, ή να καταγράψουμε, βάση περιπτώσει, τις ιδιαιτερότητες ε, του κάθε τόπου και τα εδαφικά χαρακτηριστικά, ε, αλλά και να θέσουμε προηγουμένους στόχους για μια συγκεκριμένη περίοδο, ό,τι αφορά το περιβάλλον. Έτσι, και οι τοπικές αρχές θα μπορούσαν να δράσουν καλύτερα και οι γεωργοί αλλά θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον. Ολοκληρώνοντα να πω ότι βεβαίω ε, και ε, όταν θα υποβληθούν οι τροπολογίε θα προτείνω μία ε, συνεδρίαση, συνάντηση με του χειώδει εισηγητέ και σίγουρα με στόχο την βελτίωση αυτών των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος από τους σκιώδες είναι παρόν. Ο κύριος ίσως θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια γιατί τόσο εις βάθος ανάλυση που θέλησε να μας δώσει της χρηματοδότησής της. Η πρόταση είναι ήδη ευρύτατη, πολύ καλά διαρθρωμένη σε γενικές γραμμές ασπάζομαι τις θέσεις της ηγητρίας. Παρά τα αυτά, αισθάνομαι ότι οφείλω να κάνω κάποιες σκέψεις πάνω από το πρίσμα των ενδιαφερόντων της Επιτροπής μας. Επί της αρχής να πω ότι βλέπω θετικά τη δομή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την πρόταση κανονισμού. Ιδίω σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και τη στήριξη στους νέους ερχόμενους και τις μειονεκτικές ε, περιφέρειες. Αρχή τη αλληλεγγύης, εν προκειμένου. Επίσης, ε, σκόπιμη θεωρώ ε, την εισαγωγή του καθεστώτος του πρασινίσματος, του greening Βεβαίω, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία εν προκειμένου. Ευελιξία σε ό,τι αφορά την εντατική ε, καλλιέργεια θαμνοδών ε, φυτών και της ε, αμπέλου. Ώστε να, να μπορέσουν να επιτύχουμε τους περιβαλλοντικούς τόχους που απαιτούνται. Και είναι βασικό χαρακτηριστικό του greening. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο δύσκολες είναι οι αλλαγές ε, βεβαίως ε, στις καλλιέργειες και στο φυσικό τοπίο. Ιδίως όταν μιλάμε για λόφους και για τη Νότιο Ευρώπη, ιδίως αναφέρομαι στη Μεσόγειο. Σε ό,τι αφορά την απέτηση του greening κατά 30% θεωρώ ότι το σύστημα της πολλαπλής συμμόρφωσης έχει ως σκοπό την εκπλήρωση των στόχων, ταυτόχρονα όμως δεν θέτει προσιλοποίηση και τον αντίστροφο, αν θέλετε, μηχανισμό. Δηλαδή, να μπορούν να επιτευχθούν οι μέγιστες άμεσες ενισχύσεις, διατηρώντας λοιπόν τις καλλιέργειες που επιτρέπονται πλέον στις περιοχές που μπορούν να ενταχθούν, ε, που είναι επιλέξιμες αυτούς τους στόχους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ευρύτερη γκάμα επιλογών σε ό,τι αφορά το greening, υποχρεωτικό greening μεν, αλλά επιτρέποντας να γίνουν δύο τουλάχιστον επιλογές που θα γίνονται στην ε, πρώτη φάση. Επίσης είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη, πάντοτε στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας, να έχουν τη δυνατότητα να ε, ορίζουν το καθεστώς του μικρού αγρότη, ανάλογα με τις παραδόσεις και την εθνική νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. Τέλος, σκόπιμο θα ήταν να διευρυνθούν οι διατάξεις που αφορούν τις παραμεθόριες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου και όλες οι νησιωτικές περιφέρειες που έχουν να αντιμετωπίσουν συνεχώς πολύ υψηλότερο κόστος προμήθειας τροφίμων και λοιπόν βασικών εμπορικών αγαθών, καθώς το κόστος αυτός είναι πολύ ψηλότερο του μέσου όρου για την υπηρετική Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, για το ΕΛΚ, η κυρία Τσικίσκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ φιλόδοξη αυτή η πρόταση για τις ε, άμεσες ενισχύσεις. Η συγγήτρια είπε ότι οι κείμενες προτάσεις δεν είναι αρκετά ε, ισχυρές. Βεβαίω πρέπει να χρησιμοποιηθούν πόροι για να καταλήξουμε στο να έχουμε μια γεωργία πιο φιλική στο περιβάλλον. Βεβαίω αυτό θέλουμε να υποστηρίξουμε όλοι. Όμω το περαιτέρω υψηλότερο μόνο επίπεδο πρασινίσματος, greening, ε, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα και σε ανησυχίες και φόβους μεταξύ των αγροτών. Γιατί ποιο ακριβώ θα πληρώσει το τίμημα για αυτό το greening, οι ίδιοι οι αγρότες. Να μην ξεχνάμε ότι το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα και οι άμεσε ενισχύσει δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως το δεύτερο πυλώνα, σημείο 13 της ε, έκθεσης. Και επίση η πρόταση για το 30% των κονδυλίων υποχρεωτικά να διοχετευτεί στην οικολογική γεωργία σε μειονεκτικές περιοχές. Για το δεύτερο πυλώνα όμως το 50% των κονδυλίων θα δαπανηθεί για το πρασίνισμα, αν καταλαβαίνω καλά. Άρα, ποια δεν τα κονδύλια θα απομείνουν για τις πραγματικές επενδύσεις στο δεύτερο πυλώνα, για την ε, καινοτομία, για την πρόοδο. Αυτό δηλαδή που πρέπει να χρηματοδοτήσει ο δεύτερος πυλώνας. Θα είναι πολύ λιγότερα ουσιαστικά τα κονδύλια για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου δεν θα υπάρχουν ουσιαστικά καθόλου κονδύλια για την ανάπτυξη της υπαίθρου, για τις ε, καλύτερες τεχνολογικές υποδομές, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Όλα αυτά θα πρέπει μετά να βαρύνουν την πολιτική συνοχής. Το μόνο δηλαδή που θα πρέπει να απασχολεί τους αγρότες είναι το greening, είναι το πρασίνισμα. Ε, γνωρίζοντα ταυτόχρονα ότι αυτό θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας έναντι άλλων χωρών του κόσμου. Να μην ξεχνάμε όμως ότι το ίμιση ε, του εισοδήματο του Ευρωπαίου αγρότη προέρχεται από τις ε, άμεσε πληρωμές. Άρα Βεβαίω και θα πρέπει η γεωργία να είναι φιλική προ το περιβάλλον. Δεν διαφωνεί κανένα με αυτό. Αυτό το διευκρινίζει πολύ καλά η Κομισιόν στην πρότασή τη. Έχει στηθεί το θέμα επί Μακρόν και στην Επιτροπή Άγκρη, η οποία προσπαθούσε όμω να βρει κάποιε λύσει πιο φιλικέ και ευνοϊκέ για τον ίδιο τον αγρότη. Αλλά τελικά ο τελικός προϋπολογισμός για την ΚΑΠ δεν αυξήθηκε, ουσιαστικά μειώθηκε, διότι παραμένει μεν ο ίδιος, αλλά έχουμε πιο πολλές δικαιούχες χώρες. Άρα, ουσιαστικά έχουμε περικοπή. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί κίνδυνοι, θεωρώ, από αυτές τις προτάσεις πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερη προσοχή ώστε αυτά που θα αποφασίσουμε να μπορέσουν να λειτουργήσουν στην πράξη, να είναι αποτελεσματικά. Οι συνεχείς περικοπές ε, που ψιθυρίζονται για την κοινή αγροτική πολιτική ουσιαστικά δέρνουν το δεύτερο πυλώνα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή τις θέσεις εργασίας, την προσοχή του περιβάλλοντος και όλες τις άλλες πολιτικές που ανέφερα πριν. Τώρα, η Επιτροπή προτείνει 10% να περάσει από τον πρώτο στο δεύτερο πυλόν, εμείς προτείνουμε στην έκθεση 20%. Αυτό όμως δεν είναι υποχρέωση, είναι μια δυνατότητα. Να το δούμε, δεν διαφωνώ, να το συζητήσουμε. Δεν πιστεύω ότι θα έρχεται κανένας ε, απόλυτα ικανοποιημένος από αυτό το ενδεχόμενο. Επίσης, η διαφοροποίηση των επιπέδων στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα, δείτε για παράδειγμα, τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν για την Πορτογαλία και την Πολωνία και τη Γαλλία που πάει μόνο μέχρι το 8%. Αν αλλάξουν αυτά τα ποσοστά για το δεύτερο πυλώνα, να είμαστε προσεκτικοί για τις συνέπειες που θα έχουμε. Βεβαίως υπάρχει και πρόταση να περάσουν κάποια πράγματα από το δεύτερο στον πρώτο πυλώνα. Κάτι για 12 με 15% άκουσα για κάποια κρατημέλη. Η συνάδελφος προτείνει 5%. Κατανοώ τη λογική της συγγήτριας. Όμως, με έναν ελληπή προπολογισμό, με έλλειψη κονδυλίων, αν μειώσουμε τις πληρωμές για τα νεα κρατημέλη, καποια κρατημέλη θα θέλουν να κάνουν αυτό το πέρασμα από το δεύτερο στον πρώτο πυλώνα αυτή τη μεταφορά για να μπορέσουν να ε, αντισταθμίσουν αυτό το τρόπο αυτή την αρνητική εξέλιξη. Κοιτάξτε, τρόπον την δίκιο έχει συνάδελφος σε πολλά σε όσα λέει για την βιοπικιλότητα, ε, ότι είναι πολύ σημαντικό τώρα να έχουν πιο πολλέ καλλιέργειες από λιγότερες. Ποιος διαφωνεί με κάτι τέτοιο. Όμως, οι ποικιλίε στις καλλιέργειες θα πρέπει να έχει και ένα πρακτικό νόημα, να χρησιμοποιούνται όλες τις καλλιέργειες. Πρέπει να είμαστε και λιγάκι λογικοί, ε, προσγειωμένοι στο έδαφος. συμφωνώ με την εισαγωγή ε, νέων ε, ποικιλιών. Και να ρωτήσει κανείς, γιατί εισάγουμε τόσους μεγάλους όγκους όγιας. Θα πρέπει δηλαδή οι τελικές επιλογές να είναι βιώσιμες ε, για την ευρωπαϊκή γεωργία. Έπειτα, θέλω να αναφερθώ στο 7% της γεωργικής χρήσης από τις οικολογικές υποδομές, τις λεγόμενες οικολογικές υποδομές. Σκεφτείτε όμως την εντατική καλλιέργεια, εντατική γεωργία, στην Ολλανδία π.χ. Αν αποκλειστεί το 7% αυτών των εκτάσεων, τελικά δεν θα υπάρχουν ε, ούτε δασικές εκτάσεις, ούτε άλλες εκτάσεις που συμβάλλουν στο πρασίνισμα. Αυτό το 7% λοιπόν που θα πρέπει να μην χρησιμοποιείται από τη γεωργία για το πρασίνισμα, το πώς δηλαδή υπολογίζεται, ε, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ προσεκτικοί. Πώς θα προστατεύσουμε και τη βιοπικιλότητα ταυτόχρονα. Βιοπικιλότητα και διαφύλαξη ανταγωνιστικότητα στις γεωργίες μας. Μια ευρωπαϊκή γεωργία που είναι ελάχιστα ανταγωνιστική ήδη Ο κίνδυνο είναι διάφορε αγροτικέ εκμεταλλεύσει να πάνε να εξαγοράσουν αυτό το 7% από αλλού, από άλλες χώρες. Για να μπορούν να έχουν μια τελική αρρώσιμη έκταση, ε, ε, βιώσιμη ε, οικονομικά. Ό,τι και τελικά αν επιλεγεί, εμεί συμφωνούμε το γενικό κανόνα ότι θα πρέπει η γεωργία να προστατεύει το περιβάλλον. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει εκπρόσωπο τη ΓΔ Άκρη. Παρακαλώ, θέλετε το λόγο. if you were a man, I'm, I'm terribly sorry, but I'm sorry. It's fine. I, I said Mr. <laughs> yeah, no, okay, no problem. Όμως σας είπα κύριο. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετικά εις βάθος ανάλυση για τις προτάσεις του, για το σκιώδη εισηγητή επίσης ευχαριστώ για τα σχόλια που μας παρουσίασε, τα έχω σημειώσει καθώς και τον τελευταίο ομιλητή και θα παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή τις επόμενες εβδομάδες τη συζήτηση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Ε, I don't know if Madame Grezou, Κυρία Ρέζου, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, πολύ σύντομα. Και εγώ παρακολούθησα τους ομιλητές, σκιώδης, μέλη της Επιτροπής και βεβαίως περιμένω την υποβολή τροπολογιών. Ελπίζω να πλησιάσουμε οι μεν τους δε. Η διαπραγμάτευση όμως τελικά εξαρτάται από πολλά αλλά. Ελπίζω μέσα σε όλα αυτά τα αλλά να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή κατεύθυνση προστατεύοντας ε, τη γεωργία, αλλά κυρίως την υγεία των ε, γεωργών μας, γιατί εδώ μιλάμε για αρσιτοκτόνα, εντομοκτόνα και όπως ξέρετε τα πρώτα θύματα είναι η γεωργοί. Πρόεδρος, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών σας προτείνω στις 19 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι στις 12. Αύριο. Και νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό. Θέλω να κάνω μια γενική παρατήρηση. Συνάδελφοι, είμαστε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, γνωμοδοτούμε και κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να γνωμοδοτούμε επί κάποιων θεμάτων που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Επιτροπής μας. Οι γνωμοδοτήσεις μας λοιπόν θα πρέπει να γίνονται υπό αυτή την οπτική γωνία. Περνάμε στο 24. Ο εισηγητής ε, είναι εδώ. Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρόταση κανονισμού υπό εξέταση λοιπόν πρόταση περιέχει μια σειρά προτάσεων ώστε να έχουμε μια ομοιόμορφη αποτελεσματική εφαρμογή της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η πρόταση ορίζει τη χρηματοδότηση ε, και τα ταμεία που θα διέπουν την κοινή αγροτική πολιτική. Το Ταμείο Γεωργικών Εγγύσεων που διασφαλίζει τις ε, άβας πληρωμές, το Ταμείο που χρηματοδοτεί ε, την ανάπτυξη της υπαίθρου. Επίσης προβλέπει τη χρηματοδότηση ενός συστήματος ε, παροχής συμβουλών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ώστε να χρησιμοποιούν καλές πρακτικές με στόχο τη διασφάλιση βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και απευθύνεται στις εκμεταλλεύσεις εκείνες που μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερε δυσχέρειε ως προς τη διαχείριση και τον προσανατολισμό τους στην αγορά. Τέλος, ορίζει και διαρθρώνει το σύστημα παρακολούθησης αποτελεσματικότητας της κοινή αγροτικής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα τον αντίκτυπο στην ε, αγροτική οικονομία. Η αλήθεια είναι ότι η πρόταση αυτή, όπως πολύ ορθά είπε πριν από λίγο και η πρόεδρος ε, κυρία Χιούμπνερ, είναι μια πρόταση που εκφύσεως δεν μπορεί να εστιάσει την προσοχή σου και να έχει στο επίκεντρο την ε, περιφερειακή πολιτική. Η γνωμοδότησή μου λοιπόν, στην γνωμοδότηση αυτή προσπάθησα να εντάξω μία πρόταση που εκφύσεως σίγουρα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην απέτηση του εξορθολογισμού αποτελεσματικότητας και απλούστευσης. Το να ζητήσει κανείς σημαντικές και πολλές αλλαγές στην αρχική πρόταση θα μπορούσε να κρυθεί μη σκόπιμο και να μην βοηθήσει στο τελικό σκοπό και να μην οδηγήσει στην επιβολή των στόρων ρυθμίσεων. Προσπάθησα λοιπόν να εστιάσω την προσοχή μου σε αυτή τη γνωμοδότηση σε λίγες αλλά θεωρώ καθοριστικές παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα έκρινα σκόπιμο να λειτουργήσω από το γνώμα της αλληλεγγύης και να δώσω έμφαση στη πιο, στο πιο δύναμο κρίκο της αγροτικής αλυσίδας, ώστε να υπάρχει εξορθολογισμός, χρησιμοποιώντας όσο γίνεται περισσότερο την κοινοτομία. Μία προσέγγιση που εγγυάται τα καλύτερα σε αποδυναμωμένες σήμερα αγροτικές κοινωνίες που αντιμετωπίσουν τη μείωση του πληθυσμού, ενώ η γεωργία παραμένει πηγή παράδοσης και κοινωνικού πλούτου, ίσως, αλλά και μάλλον και οικονομικού πλούτου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και άλλες αιτίες που επηρεάζουν τελικά τα αγροτικά εισοδήματα σήμερα σε τέτοιο δραματικό ρυθμό. Θα πρέπει να βοηθήσουμε για την καλύτερη διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ώστε οι πληρωμές ε, που λαμβάνουν να μπορούν να εγγραφούν ε, στον ισολογισμό των ε, αγροτικών επιχειρήσεων. Προτείνω επίσης από τη μία πλευρά αύξηση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την επιλογή των φορέων πιστοποίησης και από την άλλη να συσχετίσουμε το σύστημα περιβαλλοντικής συμβουλής με τον ακαδημαϊκό κόσμο της εκάστοτε περιοχής. Οπότε να διευκολύνουμε τις διαδικασίες ε, της ένταξης της καινοτομίας στην αγορά εργασίας και της παραγωγής. Τέλος, ό,τι αφορά την παρακολούθηση της αγροτική πολιτικής, σκόπιμο είναι να εντάξουμε μια σειρά δικτών που θα μας επιτρέψουν με αποτελεσματικό τρόπο να δούμε πώς, τι αντίκτυπο μάλλον έχει η αγροτική πολιτική σε όλες τις πτυχές του βίου. Πιο συγκεκριμένα προτείνω να εισάγουμε δείκτες σχετικά με την πρόσβαση στι αγορέ, η διαδικασία κατάρτισης, η διαδικασία διαμόρφωσης και σταθερότητα των τιμών και άλλους δείκτες ε, που να μετρούν το ποσοστό ε, χρήσης ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή. Έπειτα, δείκτες που να μπορούν να μετρήσουν την ανάπτυξη της υπαίθρου, τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο. Έπειτα, αστική κινητικότητα, δημογραφικές τάσεις και ποσοστά φτώχεια στις αγροτικές περιοχές. Να σταματήσω εδώ. Εκτός αν έχω άλλα δύο λεπτά στη διάθεσή μου, Έχω χρόνο, Πρόεδρε, διότι εγώ σας ανέφερα τώρα τις βασικές ε, τροπολογίες μου. Αλλά αν έχουμε χρόνο μπορώ να επανέλθω. Thank you very much, Sean Kelly. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Κέλλη. Ε, thank very much. Ε. Ευχαριστώ πολύ, καταρχήν. Θα ήθελα να πω ότι ευτυχώς που έχουμε συζήτηση για το θέμα αυτό, και δεν έχουμε την ίδια περίπτωση όπως με τον άλλο συγκεκτή που τελικά αποφάσισε να μην γίνει συζήτηση. Μπορούμε να υποβάλουμε και τροπολογίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για μας, διότι όλες οι περιφέρειες εξαρτώνται από τον τομέα το γεωργικό και την βιωσιμότητά του και οι στόχοι της στρατηγικής 2020 και οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται σε αυτή μας οδηγούν σε μεγάλη εξάρτηση από τον τομέα αυτό και ιδιαίτερα από τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Βλέπουμε ότι σε πολλές περιφέρειες πλήττεται ο τομέας αυτός, πλήττονται οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Γι' αυτό και αυτό που είπε ο εισηγητής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη σιγουριά οικονομική για τους γεωργούς, ότι οι πληρωμές καταβάλλονται εγκαίρος Στη χώρα μου την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε ότι κάποιες πληρωμές είχαν καθυστερήσει από τον ε, Σεπτέμβριο στον... Μάλλον κάποιες ε, πληρωμές του Δεκεμβρίου θα γίνουν το Σεπτέμβριο εξαιτίας ε, των καταστροφών μετά από τις καιρικές συνθήκες που γνώρισε η περιοχή το καλοκαίρι. Βεβαίως από εκεί και πέρα το θέμα είναι το πόσο έγκαιρα θα καταβληθούν τα ποσά και πόσο έγκαιρα θα μπορέσουν οι γεωργοί να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε τις μεταβολές στην κοινή αγροτική πολιτική, κάτι που όπως φαίνεται θα οδηγήσει μάλλον σε αύξηση και όχι σε μείωση των οικονομικών δυσκολιών που γνωρίζουν σήμερα οι αγρότες. Κάποιες αδυναμίες και κάποια σφάλματα θα πρέπει να εντοπιστούν. Το θέμα της έρευνας. Βεβαίως, θα πρέπει να στηρίξουμε ερευνητικά προγράμματα που έχουν άμεση επιπτώσεις στην γεωργία, στην ανάπτυξη και πρόθεση ποιοτική διατροφικής αλυσίδας, ποιοτικών τροφίμων. Και βεβαίως αυτό που είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή είναι και η ανάπτυξη και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων όπως ο αγροτουρισμός, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά βεβαίως κυρίως οι δραστηριότητες αυτές που έχουν σχέση με τη γεωργία Πιστεύω ότι όπως και άλλοι θα υποβάλω τροπολογίες που θα ενισχύσουν όλες αυτές τις πτυχές έτσι ώστε θα μπορέσουμε να στηρίξουμε όχι μόνο την καθαρά γεωργική δραστηριότητα αλλά και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χρυσόγελ. Σίγουρα η αγροτική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντική και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ε, η γεωργία μόνο, δεν είναι μόνο μια παραγωγική δραστηριότητα, αλλά πολλές φορές έχει συμμετάσχει και έχει συμβάλει στην πολιτισμική ανάπτυξη των περιοχών και στη διατήρηση των οικολογικών χαρακτηριστικών περιοχών. Ε, τουλάχιστον σε ορισμένες μορφές ε, αγροτικής δραστηριότητας και πρακτικές που ακολουθούνταν στο παρελθόν διαπιστώνουμε μια μεγάλη σοφία, όπως ήταν το θέμα με τις αμυσπορές ή αυτό που παρατηρούμε στον Νότο, στις περιοχές που υπήρχε μεγάλη κλίση, η δημιουργία των αναβαθμίδων, ε, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για την καλλιέργεια του εδάφους, αλλά και έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την διατήρηση των οικολογικών χαρακτηριστικών, για τον εμπλουτισμό του υπεδάφους με νερό κλπ. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους γεωργούς να προσαρμοστούν στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να επιλέξουν τις καλύτερες λύσεις και για τη γεωρική δραστηριότητα, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του κλίματος. Και ταυτόχρονα να μπορούν να έχουν εκείνες τις υποδομές σε σχέση με τη δημόσια υγεία, ε, να γνωρίζουν τα θέματα της υγείας των ζώων, ε, καινούργιες τάσεις που υπάρχουν και μεταξύ των καταναλωτών. Δηλαδή αυτά όλα νομίζω ότι είναι στοιχεία της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής και θα πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες να προσαρμοστούν και το πρασίνισμα ή και οι εκτάσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, για ε, το πρασίνισμα σε καλλιέργειες, ακόμα και μονοκαλλιέργειες, νομίζω συμβάλλουν και στην βελτίωση του εισοδήματος του ίδιου του αγρότη. Πολλές από τι ασθένειε, οφείλει σε γεγονό ότι έχουμε εκτεταμένε μονοκαλλιέργειε. Και άρα έχει χαθεί η ισορροπία στο αγροτικό περιβάλλον και αυτό έχει πολλέ φορέ επίπτωση και οικονομική, γιατί οι αγρότε είναι περισσότερο εξαρτημένοι από τα λοιπάσματα και από τα φυτοφάρμακα. Ιδιαίτερα σε μια εποχή σαν τη σημερινή, που η εξάρτησή του από ε, τι πρώτε ύλε που έρχονται έξω από το χωράφι αυξάνει τα χρέη του προ τι τράπεζε. Εάν σκεφτούμε πώ ήταν παλιά ένα γεωργό, ήταν εξαρτημένο από τη δικιά του δουλειά, ενώ σήμερα είναι εξαρτημένο πλήρω από, από την εισαγωγή ενέργεια, ε, σπόρων, ε, φυτοφαρμάκων, λοιπασμάτων κλπ. Άρα το πρασίνισμα τη γεωργίας και η έμφαση στο πρασίνισμα τη γεωργία θα βοηθήσει και τον αγρότη να έχει καλύτερο εισόδημα και να ξαναεπιστρέψει σε μια μεγαλύτερη αυτάρκεια στο περιφερειακό επίπεδο. Όμως δεν είναι εύκολη αυτή η μεταστροφή γιατί πολλές φορές έχει χαθεί η γνώση ε, αλλά και την άλλη μεριά απαιτείται σύγχρονη επιστημονική γνώση και πράγματι πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία, στην επιστημονική γνώση, αλλά και σε μηχανισμούς συμβουλευτικού προς τους αγρότες, γιατί ένα μεγάλο, έχουμε χάσει ε, εκείνο το ρόλο που έπαιζαν οι επιστήμονες στην Ήπεθρο, παράδειγμα οι γεωπόνοι, που συμβούλευαν τον αγρότη πώς να καλλιεργεί. Σήμερα οι περισσότεροι γεωπόνοι ή απλώς γράφουν συνταγές για φυτοφάρμακα ή συμπληρώνουν ε, διάφορες ε, γραφειοκρατικές ε, αιτήσει και έχουν να ανταποκριθούν περισσότερο σε γραφειοκρατικά θέματα. Στη χώρα μου, αλλά νομίζω στο Νότο ιδιαίτερα, γενικότερα, λένε πολύ συχνά ότι πλέον ο γεωπόνο δεν είναι στο χωράφι να συμβουλεύσει τον αγρότη, που είναι αυτό ο ρόλο του, αλλά είναι σε ένα γραφείο και συμπληρώνει αιτήσει και διεκπεραιώνει γραφειοκρατικέ υποθέσει. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε αυτούς τους συμβουλευτικούς θεσμούς στους αγρότες και ιδιαίτερα στους νέους αγρότες και πώς αυτές οι συμβουλές θα στηρίζονται σε επιστημονική γνώση και θα είναι προσαρμοσμένες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά περιοχών. Παράδειγμα, επειδή κατάγουμε από μια νησιωτική περιοχή, η γεωργία στα νησιά δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τη γεωργία σε ένα κάμπο ή με τη γεωργία στο, στην Ολλανδία ή τη γεωργία στο Βέλγιο είναι ακόμα και μεταξύ των νησιών υπάρχουν μεγάλες διαφοροποίησεις. Ποιος λοιπόν θα μπορέσει να βοηθήσει τον αγρότη για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις δυνατότητες που έχει ένα νησί. Και όμως υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες γιατί η κάθε περιοχή έχει διαφορετικές δυνατότητες να αναπτυχθεί ένας τομέας ο οποίος ήταν προσαρμοσμένος στα οικολογικά χαρακτηριστικά, στα ανθρώπινα και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής, αλλά σίγουρα χρειάζεται ο αγρότης σημαντική υποστήριξη. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά τους μηχανισμούς αυτούς υποστηρικτικούς ε, για τους αγρότες. Και βέβαια να λάβουμε υπόψη όταν μιλάμε για μια πολιτική, νέα κοινή πολιτική που είναι για το 2020 μέχρι το 2020 αλλά και μακροχρόνια αυτή η κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι μέσα στα επόμενα 8 χρόνια μπορεί να έχουν συντελεστεί ακόμα μεγαλύτερε αλλαγέ στο κλίμα. Άρα θα πρέπει να είναι και οι δομές οι οποίες θα υποστηρίξουν τον αγρότη σε σχέση με τις αλλαγές που γίνονται στα οικοστήματα εξαιτία του κλίματος. Και αυτό το διαπιστώνει κανείς. Αν κάποιος γυρίσει και μιλήσει με ανθρώπους που είναι γεωργοί, που ζουν στην Ήπεθρο αλλά και πολύ ο Γεωργίος, θα δείτε ότι είναι πολύ αγχωμένοι ακριβώς για το τι θα καλλιεργούν τα επόμενα χρόνια, πώς θα προσαρμόσουν τη δραστηριότητά τους στις νέες συνθήκες, παράδειγμα φέτος υπερβολική ανομβρία και με υψηλές θερμοκρασίε για πάρα πολλέ μέρε αλλάζει πλήρως. Βλέπουμε ότι υπάρχουν καταστροφές, καλλιέργειες και αυτό μπορεί να έχει και αποτέλεσμα 50% μικρότερε αποδόσεις. Άρα όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα εντάξουμε στην καθημερινότητα του αγρότη. Γιατί είναι άλλο πράγμα το συζητάμε σε επίπεδο πανεπιστημιακό, σε επίπεδο φόρουμ και άλλο πράγμα να μπορεί να είσαι δίπλα στον αγρότη και να μιλά για αυτά τα πράγματα και να του δίνει συμβουλέ τι να κάνει το αύριο, δηλαδή πώ θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και βέβαια να τελειώσω, είναι πολύ σημαντικό το θέμα της έγκαιρης πληρωμής. Αυτό δεν αφορά μόνο τους αγρότες βέβαια, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί σήμερα οι αγρότες είναι χρωμένοι στις τράπεζες. Κάθε καθυστέρηση σημαίνει ότι επιβαρύνει το κόστος της παραγωγής, γιατί πληρώνουν περισσότερα χρήματα στις τράπεζες, άρα αυξάνει, την εξάρτηση των αγροτών ε, από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και αυξάνει και το κόστος, μειώνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Άρα πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά οι μηχανισμοί και τα γραφεία, ώστε η πληρωμή να γίνεται σε γρήγορο, σε μικρό χρονικό διάστημα, να φτάνει γρήγορα στους ε, δικαιούχους και να φτάνει με ένα σωστό τρόπο ώστε να μην υπάρχει διαφθορά, να μην υπάρχει ενδιάμεση σπατάλη πόρων. Thank you. Uh, I don't know if... Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν ε, ο συνάδελφος από την Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, οι γυναίκες έχουν πάρει τη θέση όλων των αντρών από την Επιτροπή σήμερα. Συγγνώμη για τη σύγχυση. Κριστίνα Μπόκμαν ονομάζομαι από την Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Για αυτόν τον κανονισμό θέλω να σας μιλήσω, τον οποίο παρακολουθώ. Και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης. Είναι σαφές ότι ε, εξετάζεται τον κανονισμό αυτόν από την οπτική γωνία της ε, περιφερειακής πολιτικής. Σε μερικές ε, παρατηρήσεις να κάνω μόνο επί της ουσίας των τροπολογιών και των παρατηρήσεων σήμερα. Πρώτα απ' όλα, σε αρκετές τροπολογίες προτείνατε να πείτε κράτη-μέλη ή και περιφέρειες, and or regions. Λογικό βέβαια, εμείς το έχουμε βάλει έτσι γιατί ε, θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη, το αφήνουμε στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη αποφασίζουν πώς θα το διοργανώσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει περιφερειακό οργανισμό. Απλώς ε, το κάθε κράτο μέλος μετά αποφασίζει το πώ θα το εξειδικεύσει και πώ θα το κάνει πιο συγκεκριμένα. Ε, το γεγονό λοιπόν ότι ο όρο περιφέρεια δεν αναφέρει στον κανονισμό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Βεβαίω και θα το εξετάσουμε. Σχεδόν όλοι αναφερθήκατε στην σημασία της έγκαιρης ε, πληρωμής, ε, καταβόλης των πληρωμών στους γεωργούς και γιατί δεν μπορούμε να καταβάλουμε τις πληρωμές νωρίτερα ο τρόπος λειτουργίας ε, των ε, συστημάτων ελέγχου και το καθεξής, ε, αλλά και των πληρωμών για την περιφερειακή ανάπτυξη, είναι ότι γίνονται το Μάιο οι αιτήσει του τρέχοντος έτους και μετά πληρώνονται από την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και μετά. Αυτό σημαίνει όμως ότι το επόμενο δημοσιονομικό έτος μας αφορά για τη γεωργία. Γιατί ότι στις 16 Οκτωβρίου ξεκινά το οικονομικό μας έτος. Επομένως, το τον ένα χρόνο γίνονται οι αιτήσει και οι πληρωμές καταβάλλονται στο... τον επόμενο. Περίπου 37 δις ευρώ καταβάλλονται κάθε χρόνο σε άμεσες πληρωμές. Ε, βεβαίως θα είχε επιπτώσεις στο να μεταφέρουμε το οικονομικό έτος, αλλά ε, από τις 16 Οκτωβρίου και μετά, γιατί τότε ξεκινάμε το οικονομικό έτος, έχουμε χρόνο να κάνουμε και διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Έχουμε και τις ε, ε, προκαταβολές ή τις ε, πρώτερες καταβολές, αλλά αυτό γίνεται κατόπιν της ολοκλήρωσης των ελέγχων. Στην πρόταση που έχουμε εδώ σήμερα για την επόμενη περίοδο προτείνουμε γενικές προκαταβολές κάθε χρόνο από τις 16 Οκτωβρίου και μετά. Και χαιρετίζουμε την στήριξη της Επιτροπής σας για το 42.2 που προτείναμε ε, να καταβάλλονται τόκοι από τα κράτη-μέλη ε, σε γεωργούς ε, που λαμβάνουν τις πληρωμές τους μετά τον Ιούνιο για να μην υπάρχουν και καθυστερήσει παρατέρων. Και αυτό το έχετε κοιτάξει, όμως είναι σημαντικό και για μας. Ευχαριστώ. I, I Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο Τζομαρία θέλει να απαντήσει. Δεν χρειάζεται. Μα όχι, Πρόεδρε, μόνο για να ευχαριστήσω τους, ε, τους και όσους ε, πήραν το λόγο, όπως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα όσα ακούστηκαν είναι πολύ χρήσιμα για να αποφύγουμε σφάλματα. Μόνο το εξή να αναφερθώ στο γεγονό ότι λέμε κράτη-μέλη ή περιφέρεια. Ναι, μα θεωρούμε ότι υπάρχουν διαφορετικέ αρμοδιότητε ανάλογα με τι προβλέπει η εκάστοτε ταξία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτόνομε περιφερειε σε κάποιε χώρε, κάποια συντάγματα προβλέπουν αρμοδιότητε, σε κάποιε άλλε χώρε όχι. Θα, θα τη βρούμε τη λύση βεβαίω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει διαφωνία. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να περάσει ένα μήνυμα. Το είπε και ο κύριο Κέλλη πριν λίγο ας μην εκπλαγούμε αν καταφέραμε τελικά να ο ευρωπαϊκός προπολογισμός, αν θέλετε, από τις 16 Οκτωβρίου με τη νέα δηλαδή αγροτική χρονιά να μπορέσουμε να συμπέσουμε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αγροτικού εισοδήματος. Ας ελπίσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Θα είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Η προθεσμία είναι 21 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι 12 η ώρα. Πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο θέμα επί της ουσίας, το σημείο 25, θα σας ενημερώσω για τις αποφάσεις των πολιτικών συντονιστών χθες ε, το απόγευμα αποφασίσαμε για την κατανομή εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων. Έξι γνωμοδοτήσεις για τον προπολογισμό που συνδέονται με το Ταμείο Πακοσμιοποίησης και λόγω του περιορισμού του χρόνου συνεχώς συμφωνήσαμε να μην υπάρχουν προβλήματα, θα, ε, θα αποσταλεί επιστολή του Προέδρου στην Επιτροπή Προπολογισμού ζητώντα ε, συμφωνία για έξι παραπομπές. Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία και Γαλλία. Για τις μη νομοθετικές γνωμοδοτήσεις, δύο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, συμφωνήσαμε το ΕΛΚ και οι Σοσιαλιστές Δημοκράτες να πάρουν από μία γνωμοδότηση Δεν γνωρίζουμε όμως τον εισηγητή της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Όταν δηλαδή γνωρίζουμε από ποια πολιτική ομάδα θα είναι, τότε θα αποφασίσουμε κι εμείς ανάλογα για το ΕΛΚΕ και τους σοσιαλιστές στη δική μας ε, Επιτροπή. Ποιος θα πάρει ποια γνωμοδότηση. Για την ανανεώσιμη ενέργεια τι αγορέ ενέργεια, δόθηκε στου φιλελευθέρου για τη διακυβέρνηση τη τουρκική αγορά ε, στο ECR σε ό,τι αφορά τις αντιπροσωπείες και τις δημόσιες ακροάσεις, αποφασίσαμε αρκετά γρήγορα για τις αντιπροσωπείες επόμενης χρονιάς. Έξι προτάσεις προέρχονται από το ΕΛΚ για Βουλγαρία, Βερολίνο, Σοσιαλιστές Δημοκράτες για τη Βόρεια Σουηδία και το κοσίσε στην ε, Ανατολική Σλοβακία. Οι πράσινοι πρότειναν την Κορσική και η Σαρδινία και η Γκούε προτείνει την Λαρεουνιόν. Συμφωνήσαμε ότι θα είναι τρεις ε, οι αποστολές και θα αποφασιστεί με πλειοψηφία μέσω γραπτής διαδικασίας. Θα το δούμε λοιπόν στι επόμενε ημέρε. Γιατί τις δημόσια Κροάσεις αποφασίστηκε τρει ε, δημόσια ακροασει να διοργανώσουμε το 2013. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι οι συντονιστές θα αποστείλουν στη γραμματεία την πρόταση έως τα τέλη της εβδομάδας με ε, σχετική αιτιολόγηση και στόχους. Οι τρεις ε, ακροάσεις θα αποφασιστούν και πάλι με γραπτή διαδικασία για την αποστολή στην Ιρλανδία που θα λάβει χώρα 28-29 Νοεμβρίου. Έχουμε 7 θέσεις έως τώρα, 5 υποψήφιους, ο κ. Βανίστερόι, Κρέλ, Μανέσκου, Αλφονσί και ένα μέλος της ΓΚΟΕ, δεν γνωρίζουμε ποιος ακόμη. Εξωτερικές μελέτες. Ανάθεση λοιπόν των μελετών αποφασίστηκε από τους συντονιστές να επιλέξουμε τα θέματα τη δημογραφική αλλαγή στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, το ίντερνετ και οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών και ανάλυση των συνοποιών της οικονομικής κρίσης στην κοινωνική και οικονομική συνοχή. Αυτές ήταν οι αποφάσεις των συντονιστών. Ας περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης ο κύριος Κοστολίνο είναι εδώ παρόν. Ωραία, παρακαλώ να πάρετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Είναι η δεύτερη συνάντηση με θέμα την ε, αστική πολιτική. 21 του μηνός είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, οπότε και για λόγους χρονικούς θέλω να κάνω κάποιες πρώτες σκέψεις. Πρώτα απ' όλα να πω ότι προτείνουμε για μια ακόμη φορά το εξής ε, θέμα. Ευρωπαϊκή Ένωση και αστική αναβάθμιση. Θέλουμε πιο ισχυρή ε, νομική βάση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια ευρωπαϊκή αστική πολιτική και μια ευρωπαϊκή στρατηγική πάντοτε τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας. Δεύτερη θεματική ενότητα που θέλουμε να θέσουμε είναι η διάσταση. Δεν μιλάμε μόνο για ένα αστικό κέντρο, για μια αγροτική περιοχή ως χωριστά, ε, χωριστές οντότητες, αλλά ε, να το δούμε ως σύνολο. Ένα σύνολο ε, στρατηγικό, αν θέλετε, για να υπάρχει μια ισορροπία. Από τη μία έχουμε την υπερβολική κατανάλωση, κατανάλωση πόρων στις αγροτικές περιοχές και από την άλλη αναγκαιότητα για μεγαλύτερη ποιότητα στα αστικά κέντρα. Κέντρα α, επαναχρησιμοποίησης και επαναγέννησης ε, υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου έπειτα το άστε ως η καλύτερη, το, καλύτερο, το καλύτερο μόρφωμα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ε, ενεργειακή κατανάλωση, ε, θέματα που αφορούν το κλίμα, ε, θέματα που μας απασχολούν πάντοτε, από την παραγωγή ως την καταστροφή των αποβλήτων. Ένα βασικό και κέριο ζήτημα που μας απασχολεί όλο και περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα και βεβαίως πάντοτε το μεγάλο θέμα της κοινωνικής βιωσιμότητας στις πόλεις και για τις πόλεις και όχι πλέον ε, πια στην Ήπεθρο ε, είναι που μετρούμε ακριβώς ε, την κοινωνική βιωσιμότητα, τον κοινωνικό ιστό, πώς εξελίσσεται και το θέμα της νέας φτώχειας και των νέων φτωχών στην Ευρώπη μετράται κατά κύριο λόγο στα αστικά κέντρα. Τελευταίο και μείζονο ζήτημα. Πώς θα επαναπροσανατολίσουμε την πολιτική συνοχή προς ε, την ε, αστική διάσταση και πώς τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες ε, θα εμπλακούν σε αυτό. Η πολιτική συνοχή στα επόμενα χρόνια με τον επαναπραγματισμό των πόρων για την περίοδο 2014-2020 η μεγαλύτερη προσοχή που πρέπει να προσδοθεί στα αστικά κέντρα είναι καθοριστικού και στρατηγικού χαρακτήρα απόφαση. Αλλά και για να μπορούν να δοθούν περισσότερες ε, δημόσιες ε, επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα με μια πολιτική με στόχο την ανάπτυξη. Θέλουμε δηλαδή όχι απλά ένα επιχειρησιακό περιφερειακό σχέδιο, αλλά στρατηγικά κοινά σχέδια που να αγκαλιάζουν και το Άστι και την Ήπεθρο. Για να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα κονδύλια τη πολιτική ενοχή. Τέλο, η αστική διάσταση ω κοινό αγαθό. Η ανάγκη με την πολιτική συνοχή, με την επιλεκτική ε, χρήση και τη διαφανή χρήση αυτών των πόρων καθιστά πολύ πιο πλούσια και σημαντική τη συμμετοχή του πολίτη. Η αστική λοιπόν διάσταση αυτής της προσέγγισης μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε και ένα δημοκρατικό έλλειμμα, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Κάτι πολύ σημαντικό και πολιτική συνοχή θεωρώ ότι αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της γνωμοδότησης συζητήσεις που είχα έως τώρα με τους Κιώδες και πιστεύω σε αυτό το δεύτερο γύρο συζήτησης και με το ραντεβού που θα έχουμε για την υποβολή τροπολογιών στις 21 του μήνος να καταλήξουμε σε κάτι πολύ θετικό. Παρακαλώ. Ε, thank you ε, Ευχαριστούμε πολύ. Είναι κανείς εδώ από τους Κιώδες συζητητές. Όχι. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Είναι μια ενδιαφέρουσα έκθεση και νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι αντιμετωπίζουμε τον αστικό χώρο όχι απλώς ως ε, κτίρια, ως ε, θέματα ενέργειας ή ως θέμα φυσικών πόρων, αλλά και ως ένα χώρο που ε, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι, θέσεις, οι σχέσεις των ανθρώπων και ακόμα και φαινόμενα όπως είναι το θέμα της μετανάστευσης αλλάζουν πάρα πολύ το χώρο και βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν κενά στην οργάνωση του χώρου, όταν υπάρχουν κενά στην πολιτική, τότε έρχονται ακραίε ε, πολιτικές δυνάμεις να εκμεταλλευτούν αυτά τα κενά, κάτι που συμβαίνει ιδιαίτερα σήμερα σε πόλεις και σε χώρες που υπάρχει έντονη και βαθιά κρίση. Άρα πρέπει να και η περιφερειακή πολιτική και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να δώσουν πολύ μεγάλη έμφαση και μέσα στην, στη συνολική λειτουργία της πόλης και το θέμα της συνοχής μέσα στην ίδια την πόλη ε, της, ε, να αντιμετωπίσει τα κενά που δημιουργούνται σε αυτό που η εισηγητής ονόμασε κοινωνική βιωσιμότητα ε, και από την άλλη μεριά να βοηθήσει και τη σχέση μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου σε μια πιο υγιή βάση. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη σημερινή εποχή της κρίσης σε δύο σημεία τα οποία τόνισε και ο μιλ... μάλλον σε ένα σημείο που τόνισε ο μιλητής, στη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της πόλης. Ε, και ας μην ξεχνάμε ότι μέσα στις πόλεις γεννήθηκε και η δημοκρατία και ο πολιτισμός. Ορισμένες πόλεις σήμερα είναι σε φάση αναγέννησης και ανάπτυξης με την ευρύτερη έννοια. Ε, υπάρχουν όμως άλλες πόλεις που πέφτουν σε βαθιά κρίση και χάνουν και τα στοιχεία της συμμετοχή και τα στοιχεία της δημοκρατίας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση, είναι πολύ σημαντική η προσέγγιση αυτή που υπάρχει και στην έκθεση, και ε, θα καταθέσουμε και παρατηρήσεις και προσθήκες ε, στην, ε, στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Uh, παρατηρήσεις από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής. Θα, ήθελα, θα θέλαμε να χαιρετήσουμε την ε, συζήτηση αυτή που ξεκινά από την ε, έκθεση του εισηγητή ε, για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Μερικές παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω για κάποια από τα σημεία της έκθεσης. Η Επιτροπή πράγματι έχει προτείνει την ενίσχυση της ε, αστικής ανάπτυξης μέσω της, ε, ε, της πολιτικής συνοχής με αφιέρωση του 5% του Ταμείου για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Στην έκθεση αναφέρεται... Γίνεται άμεσα αναφορά στις ε, τοπικές αρχές. Εμείς αναθέτουμε τη διαχείριση αυτού του, του 5% ε, στις ε, αστικές αρχές. Πάμε να δούμε παραπέρα λοιπόν. Άλλη αναφορά γινόταν στην πλατφόρμα αστικής ανάπτυξης. με στόχο την αναφορά στην επέκταση στις αστικές περιοχές δηλαδή και στις πόλεις και στις αστικές περιοχές. Θέλετε να επανέλθετε. Κοιτάξτε, είναι τόσο περίπλοκο αυτό το ζήτημα που δεν μας στάνει αυτός ο Απλά θέλω να επισημάνω το εξή σε όλους μας και στην Κομισιόν. Οι προβολές για τι επόμενα 30-40 χρόνια λένε ότι οι, τα μεγάλα μετροπολιτικά κέντρα και οι διαστάσεις που θα πάρουν θα έχουν καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές ανάπτυξης. Ήδη στην Ευρώπη αυτό συμβαίνει. Ήδη το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ παράγεται στα αστικά κέντρα πολύ μεγάλο μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε αφορούν και βρίσκονται στα αστικά κέντρα. Άρα, το να πρικίσουμε την Ευρώπη, αν θέλετε, μέσω προσαρμογής πολιτικής συνοχής, μια στρατηγικής ε, πολιτικής σχετικά με τα αστικά κέντρα, θεωρώ ότι είναι στρατηγική επιλογή για το μέλλον μας. Όχι μόνο υπό την κλασική έννοια του όρου, αστικά κέντρα, υπέτρους λοιπά, αλλά υπό νέους όρους. Και ποια είναι αυτή η νέα διάσταση που εννοώ. Πρέπει να δούμε τα αστικά κέντρα με άλλα μάτια. Δεν είναι το άστια έναντι της υπαίθρου. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μια μεγάλη ε, διάκριση ανάμεσα στην προστασία της υπαίθρου, της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι η ύπεθρος, ε, η παράδοση αλλά και από την άλλη προστασία των ιστορικών πόλεων, των ιστορικών κέντρων, των αστικών κέντρων. Είναι πάντοτε αυτοί οι δύο πυλώνες. Η Κομισιόν προτείνει αυτό το 5%, προτείνει αυτή την κατεύθυνση, αυτή την προσέγγιση, πολύ ωραία, συμφωνώ. Αλλά ας φανούμε λίγο πιο φιλόδοξοι, ας ανεβάσουμε τον πύχη λίγο πιο πάνω. Θεωρώ ότι εδώ μπορούμε να χαράξουμε μια καλύτερη πολιτική ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη ευχαριστούμε πολύ. Καταληκτική ημερομηνία είναι 20 Σεπτεμβρίου ε, στις 12 το μεσημέρι. Και η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 8 Οκτωβρίου. Θα επικεντρωθούμε στη... σε αυτό το Open Days. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. φορές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 Μακόγα Sinan.